Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι ήδη 9 και 10 και νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. Να σας πω ότι θα ξεκινήσουμε με το σημείο 11 της ημερησίας διατάξεως που αφορά την συνέχιση ανταλλαγή απόψεων ε, με τον κύριο Ιωάννης Χάν, Επίτροπο Αρμόδιο για Περιφερειακή Πολιτική δεν είχαμε χρόνο την προηγούμενη φορά και είπαμε ότι οι συνάδελφοι που είχαν εγγραφεί ήδη στη λίστα των αγορητών θα μπορούσαν να πάρουν τον λόγο σήμερα. Να σας υπενθυμίσω επίσης ότι έχουμε και τον κύριο Αγκουρακά και τον κύριο Ζέμπερ, τον κύριο Ματούλα, τον κύριο Βάουνς, Κότα, Σίμον και Όμπερ Μάιερ. Αυτή είναι η από την προηγούμενη φορά και όσοι θέλουν, ο κύριος Αγκουράκης δεν είναι εδώ, εν πάση περιπτώσει Όποιο θέλει να μιλήσει, να γραφτεί στον κατάλογο και βεβαίω να είσαστε λακωνικοί και συγκεκριμένοι στι ερωτήσεις Ο επίτροπο συμφώνησε να μην μιλήσει ε, σε, καταρχήν. Ζέμπερ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Χαίρομαι που τηρείται αυτή η υπόσχεση η οποία εδόθηκε την τελευταία φορά. Τρία ερωτήματα στον κύριο Επίτροπο. Κύριε Επίτροπε, πώς βλέπετε το θέμα του mainstreaming, της, της περιφερειακής πολιτικής μετά το 2013 υπάρχει αίτηση πάρα πολλών επιτροπών να υποστηριχθούν προγράμματα στον τομέα της ε, κλιματικής αλλαγής. Ε, πώς ε, θεωρείτε ότι μπορεί να αντιμετωπιστεί το σύνολο αυτών των αιτήσεων που έχουν να κάνουν με την ε, Περιφερειακή Επιτροπή. Δεύτερον, στην Επιτροπή Περιβάλλοντος η έκθεση GDB δεν έγινε δεκτή γιατί κατά την άποψή μα περιλάμβανε πάρα πολλού παράγοντε οι οποίοι δεν ήταν μετρήσιμου χαρακτήρα. Ποια είναι τα μέτρα τα οποία εσεί θέλετε να προτείνετε ώστε να μπορέσουμε στο μέλλον να επιτύχουμε την υποστήριξη των καταλήλων προγραμμάτων. Τι προτείνετε λοιπόν από τη δική σα πλευρά και τρίτον, χθε ε, την επιτροπή μα ήταν ο κύριο Ροσμπάχερ, ο οποίο είναι γνωστό σε εσά από την Αυστρία και ο οποίο είχε πει μεταξύ άλλων ότι τα ε, μπερδεμένα προγράμματα, τα πολύπλοκα προγράμματα δημιουργούν προβλήματα για τους Αυστριακούς και τι τις δομέ. Και το ερώτημα είναι αν τα συστήματα που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ήδη πάρα πολύ πολύπλοκα ή όχι. Ευχαριστώ. Δεν είναι εδώ ο Σαντφός Σωματούλα.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 για το θέμα της εφαρμογής και ίσως είναι θέματα απλώς κατανόησης. Εγώ καταλαβαίνω την ερεσιμότητα και τα κίνητρα ότι μπορεί κανείς να έχει καλύτερη χρηματοδότηση αν τους στόχους οι οποίοι έχουν τεθεί προηγουμένως τους έχει ξεπεράσει, όχι απλώς εκπληρώσει. Αλλά αυτός, αυτό δημιουργεί σε ένα κίνδυνο ότι οι αποδέκτες των χρημάτων θα ε, υποτιμούν καταρχήν τους δείκτες που πρέπει να επιτευχθούν και μετά στη συνέχεια θα δείχνουν ότι τους έχουν ξεπεράσει. Αναρωτιέμαι λοιπόν στο, στην πράξη αν θα πρέπει να υπάρξει κάποια προσεκτική εξέταση για την χρησιμοποίηση των ποσών αυτών, τα οποία δεν έχουν, ε, δεν έχουν εκταμιευτεί προηγουμένως, προτού δοθούν πρόσθετα χρήματα μέσα στα πλαίσια αυτής της διαδικασίας. Θα κλείσουμε αυτή τη διαδικασία και μετά θα ακούσουμε τους συντονιστές. Σας ευχαριστώ για τον κύριο Ζέμπα. Ο στόχος μας και το προκείμενο στις συζητήσεις με τα κράτη-μέλη ήταν να μπορέσουμε από τη βάση ουσιαστικών διαπιστώσεων όπου εμπλέκονται φυσικά όχι μόνο οι αρμόδιοι της ε, περιφερειακής πολιτικής αλλά και εκπρόσωποι άλλων πολιτικών οι οποίοι <coughs> είχαν προσκληθεί ε, ήταν παρούσες διάφορες ε, εκπρόσωποι από task force στον τομέα της ενέργειας της κλιματικής αλλαγής δηλαδή όλες οι υπηρεσίες αυτές οι οποίες αντιμετωπίζουν κάποια θέματα υπό φακέλους να παίξουν ρόλο στην προετοιμασία η οποία θα λάβει η χώρα μαζί με τα κράτη-μέλη. Ο στόχος μας είναι από το 2012 μέσα από άτυπες συνομιλίες και διαβουλεύσεις και από το 2013 και επέκεινα μέσα από επίσημες συζητήσεις με τα κράτη-μέλη να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Ο στόχος μας είναι όσο το δυνατό είναι ταχύτερο να συντάξουμε αυτές τις συμβάσεις εταιρικής σχέσης και επενδύσεων με το κάθε κράτος μέλος που να περιέχει μια συμφωνία για το τι θα κάνει το κάθε κράτος στην στις επιμέρους περιφέρειές τους και φυσικά θα περιλαμβάνει και όλες τις ρήτρες οι οποίες περιέχονται στη συνταγματική τάξη ε, αυτού του κράτους και το θέμα που θέτεται είναι ποια είναι η στοχοθεσία από τη δική μας πλευρά. Οι στόχοι μας θα πρέπει να προσαρμοστούν στη στρατηγική Ευρώπη 2020. Εκεί βρίσκονται οι προτεραιότητές μας και είμαστε πεπισμένοι ότι σε ό,τι αφορά τις περιοχές του στόχου της ανταγωνιστικότητας θα πρέπει να επιλεγούν μονάχα λίγες προτεραιότητες <clears throat> ώστε να υπάρχει στοχευμένη και συγκεντρωμένη χρήση των πόρων. Αυτό επομένως εναπόκειται στις περιφέρειες αυτές ή στα κρατήδια των κρατών μελών για να παρουσιάσουν τις πρωτοβουλίες, τις πρωτοβουλίες ή τις προτεραιότητες που θα έχουν. Επομένως, ο στόχος μας θα είναι τα, οι δομές αυτές οι περιφερειακές να επιλέξουν αυτό το οποίο θα έχει τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα για τους ίδιους τους, τους πολίτες και να μην υπάρξει ένας κατακερματισμός των κονδυλίων. Νομίζω ότι αυτό είναι ένα δρόμο ο οποίο έχει καταδείξει την αξία του στο παρελθόν, το να μπορούμε να συζητούμε με τα κράτη-μέλη, με τι περιφέρειες για τις προτεραιότητες τις οποίες θα έχουν επιλέξει τα ίδια αυτά, τα, αυτές οι ίδιες οι δομές και επί τη βάση αυτών των προτεραιοτήτων να μπορέσουμε να θεσπίσουμε στόχους οι οποίοι είναι φιλόδοξοι και ε, ποσοτικοποιήσιμοι και οι οποίοι μπορούν να υπόκεινται σε μια διαδικασία καταμέτρησης αλλά βέβαια επί τη βάση μιας ε, συμφωνίας για το πώς καταλήγουμε στα αριθμητικά αυτά στοιχεία που είναι η βάση της καταμέτρησης της επιτυχίας. Οι λεγόμενοι outcome indicators υπάρχουν ήδη και με τις ε, προσπάθειες του Φαμπρίσιο Μπάτκα, ο οποίος ήταν επικεφαλής μιας αρμόδιας ομάδος <clears throat> εργασίας, υπήρξε μια σειρά από προτάσεις για μετρήσιμους δείκτες outcome, όπως λέμε, ώστε να μπορέσουν αυτοί οι δείκτες να χρησιμοποιηθούν στις συζητήσει με τα κράτη-μέλη για να υπάρξει μια σαφής βάση επί τη οποία θα μπορέσει να γίνει στη συνέχεια η βαθμολόγηση και η αξιολόγηση της επιτυχίας που έχει επιτευχθεί στα προγράμματα αυτά με μια ποσοτικά μετρήσιμη βάση πάντα. Σε όλη αυτή την προβληματική μπαίνει και το θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και της ενεργειακής απόδυσης Βέβαια, η κάθε Γενική Διεύθυνση στην Κομισιόν θεωρεί ότι ο δικός της τομέας είναι περίπου απαράγραπτος, ότι πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθεί. Και εμείς θέλουμε εδώ πέρα να τονίσουμε ότι δεν πρέπει να υπερφορτώσουμε τη βάρκα και το σύστημα, αλλά θα πρέπει να το απλοποιήσουμε. Θα πρέπει ο στόχος μας είναι να έχουμε μια στόχοδεσία η οποία να είναι σαφής αν θέλουμε δηλαδή να διατηρήσουμε την ενεργειακή απόδοση ή όχι σε ένα πρόγραμμα, αυτό πρέπει να είναι σαφές και όχι νεφελώδες. Δική μου λοιπόν κατανόηση και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να το κάνουμε πραγματικότητα είναι ότι αυτές οι σαφείς συμφωνίες με τα κράτη-μέλη και με τις επιμέρους περιφέρειες οι οποίες περιέχουν τα αποτελέσματα τα οποία επιζητούμε να επιτύχουμε θα οδηγήσουν σε σαφείς κατευθυντήρες γραμμές από τους διαχειριστές των προγραμμάτων βάσει των οποίων μπορεί να γίνει η αξιολόγηση των προτιμωμένων προγραμμάτων και επομένω η έγκριση ή η απόρριψή του. Δηλαδή να έχουν σαφεί κατευθυντήρε γραμμέ για να κατανοήσουν κατά πόσο συνάδουν αυτά τα σχέδια και προγράμματα με τι κατευθυντήρε γραμμέ και τη στοχοθεσία που έχουμε δημιουργήσει. Έτσι ελπίζουμε ότι θα βελτιωθεί και η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των ενεργειών μας. Και σε όλους τους αυστριακούς συναδέλφους που είναι παρόντες, θέλω να πω ότι κάνω μια έκκληση σε όλους τους εμπλεκομένους, όχι μονάχα σε εσά και σε μένα, αλλά και στα κράτη-μέλη και τις ε, περιφέρειες, να κάνουν ό,τι μπορούν για να μειώσουν τη γραφειοκρατία. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Έχουμε δει πως ε, δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα, τα προβλήματα στο παρελθόν και κάνουμε τροποποιήσεις <clears throat> στις, ε, στους κανόνες μας και στην νομοθεσία μας με στόχο την ε, απλοποίηση, αλλά πολλές φορές δεν εφαρμόστηκαν αυτά στα κράτη-μέλη γιατί η τοπική νομοθεσία δεν επέτρεπε κάτι τέτοιο και αυτό είναι ένα θέμα για το οποίο πρέπει να, το οποίο πρέπει να εξεταστεί να είναι ένα από τα αντικείμενα των συζητήσεων με τα κράτη-μέλη όταν φτάσουμε στο θέμα της ερεσιμότητας. Εγώ φυσικά θέλω να μιλήσω για την έννοια του παράγοντα επιτυχίας, του success factor και η έρεσιμοτητα να έχει αυτό το πιο συγκεκριμένο χαρακτήρα ότι υπάρχουν κάποιες συμφωνίες οι οποίες πρέπει να τηρηθούν ώστε να απελευθερωθούν τα αντίστοιχα ποσά. Όλοι ξέρετε από τη δική σας χώρα, από τη δική σας εκλογική περιφέρεια, ότι υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι για τους οποίους πολλές φορές τα σχέδια και τα προγράμματα καθυστερούν να εφαρμοστούν. Εμείς έχουμε μία ευρύτερη, αν θέλετε, επισκόπηση στους τομείς ενέργειας, ε, περιβάλλοντος, μεταφορών. Και μπορώ να πω ότι στις λιγότερες περιπτώσεις είναι πρωτογενούς χαρακτήρα οικονομικού χαρακτήρα μάλλον προβλήματα αυτά τα οποία καθυστερούν την εφαρμογή, τις περισσότερες φορές είναι προβλήματα διοικητικής ικανότητος, μη μεταγραφής ευρωπαϊκών νομοθετημάτων, έλλειψη γνώσεων, ε, αδυναμία εφαρμογής πολιετών πολυπλόκων προγραμμάτων. Υπάρχουν λοιπόν πολλά τέτοια προσκόμματα αυτού του είδους και ο στόχος αυτής της αντιμετώπισης επί τη βάση της ερωσιμότητας είναι να υπάρχει μια καλύτερα προσαρμοσμένη προσέγγιση σε κάθε κράτος μέλος και σε κάθε περιφέρεια επί τη βάση των ε, ιδιαιτεροτήτων του. Αυτό μόνο να το συμφωνήσουμε φυσικά με τους εμπλεκομένους μπορούμε να το κάνουμε, δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε. Ο στόχος είναι να διευκολύνουμε και να επιταχύνουμε τις διαδικασίες. αν έχουμε ένα κράτος ε, μέλος χάρη, στο οποίο δεν υπάρχει ακόμα κτηματολόγιο και δεν ξέρουμε ποιο αγροτεμάχιο ανήκει σε ποιον, αυτό καταλαβαίνετε ότι μπορεί να σα οδηγήσει σε καθυστερήσεις. Σαν παράδειγμα. Οπότε εδώ δεν μας ενδιαφέρει το να ανταμείψουμε τους καλούς ή να κολλάσουμε τους κακούς, αλλά κυρίως να είμαστε αποτελεσματικοί. Και έρχομαι τώρα στη δεύτερη παρατήρηση. Ε, αυτού του μπόνους που δίνεται σε, επί τη βάση της απόδοσης του λεγόμενου performance reserve εμείς θεωρούμε ότι αυτό θα πρέπει να δίδεται σε περιπτώσεις που <clears throat> δεν ξέρουμε εκ των προτέρων ποια κονδύλια θα χρησιμοποιηθούν εμείς θέλουμε αυτό το υπόδειγμα να αρχίσουμε να το χρησιμοποιούμε ώστε να υπάρχει αυτό το ποσοστό μπόνους της τάξης του 10% ε, από ό,τι θεωρούμε αυτή τη στιγμή για τις περιφέρειες οι οποίες έχουν ξεπεράσει τα προβλεπόμενα. Έχουν επιτύχει μια απόδοση η οποία ξεπερνάει αυτό που έχει προβληθεί και αυτό θα είναι ένα κίνητρο πιστεύω για να υπάρχει πραγματικά αποδοτική αντιμετώπιση. Ευχαριστούμε πολύ κύριο Λάμπερ Βανίστεροι. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ σύντομα σχετικά με το, τα πρώτα που αναφέρατε. πριν από το τέλος του προηγούμενου χρόνου σε μια ολομέλεια είχαμε θίξει ορισμένα ζητήματα τα οποία ε, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικά για την εργασία μας και γι' αυτό ακριβώς θα ήθελα να τα επαναλάβω, να τα θίξω ξανά. Είναι σημαντικά και για την εργασία μας αλλά και για, την, για τον καθορισμό των προτεραιοτήτων της Επιτροπής. Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες ε, περισσότερο σαφείς πληροφορίες ε, ε, σχετικά ε, με τους τομείς της στρατηγικής 2020 και επίσης θα μπορούσατε να μας δώσετε το, ένα χρονοδιάγραμμα το, των προβλεπόμενες ημερομηνίε λοιπόν για την έγκριση των τομέων αυτών. Επίσης, πώς βλέπετε το ενδεχόμενο ή την δυνατότητα υλοποίησης ε, σε περιφερειακό τοπικό επίπεδο ε, των προγραμμάτων μας έτσι ώστε να δώσουμε μια προώθηση των ε, τοπικών περιφερειακών συμφωνιών έτσι ώστε δηλαδή να ληφθούν συγκεκριμένα, να αναλυθούν συγκεκριμένα δεσμευτικά προγράμματα σε τοπικό επίπεδο. Επίσης, την άποψή σας για την ιδέα του Φάντεν Μπραντ. Και τέλος, Έχετε κάποια ιδέα για την προετοιμασία των στρατηγικών 2020 για το κατά πόσον επομένως στην υλοποίηση της στρατηγικής και των προγραμμάτων 2020 έχουν εμπλακεί οι περιφέρειες γιατί μία από τις ελλείψεις της στρατηγικής της Λισαβόνας ήταν ακριβώς αυτό και φοβούμαι ότι επαναλαμβάνεται η ίδια κατάσταση. Δηλαδή έχουμε ένα θεωρητικό έγγραφο το οποίο όμως δεν αναφέρει συγκεκριμένα δεσμευτικά στοιχεία. Στο Κοινοβούλιο εμείς έχουμε εκπονήσει πολλά ψηφίσματα σχετικά ε, με το πώς θα πρέπει να υλοποιηθούν τα προγράμματα αυτά. Παρακαλώ. Είναι κάπως αλληλένδετα όλα αυτά τα ερωτήματα. Εμείς έχουμε προβλέψει ένα σύνολο γενικών κανονισμών που στο βαθμό του δυνατού καλύπτουν στο ευρύτερο δυνατό επίπεδο και το περιφερειακό και το κοινωνικό και το Ταμείο Συνοχής και καλύπτουν τις ανάγκες τους. Και μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει μια ιδιαιτερότητα θα πρέπει να υπάρχουν επιπλέον ιδιαίτερες ρήτρε. Επομένως, αυτό το οποίο προβλέπετε και βρίσκεται ακόμα σε συζήτηση μεταξύ μας και συνδέεται με το ερώτημα το οποίο θέσατε, το να υπάρχει ένας κανονισμός σε σχέση με την λεγόμενη εδαφική συνεργασία. ουσιαστικά μια καλύτερη, να υπάρχει μια καλύτερη ορατότητα του συστήματος και αυτό βέβαια μπορεί να μην είναι απόλυτα, <clears throat> απόλυτα συνδεδεμένο με το προηγούμενο που αναφέρατε, αλλά σε χρονικό επίπεδο επίκειται αυτή τη στιγμή <clears throat> μια αναθεώρηση των κανονισμών για τα για τα διάφορα ταμεία, το Ταμείο Συνοχής, παραδείγματος χάρη, και εγώ πιστεύω ότι επί τη βάση αυτής της αντιμετώπισης θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και σε μια περαιτέρω εξέλιξη των κανονισμών. Ο στόχος μας πάντα να έχουμε μέχρι έξι κανονισμούς σε αυτή την περίπτωση, υπάρχουν και ορισμένοι, εγώ δεν είμαι μεταξύ αυτών που έχουν αυτή την αντιμετώπιση, ότι το Περιφερειακό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από κοινού με ένα μονάχα κανονισμό. Αυτό όμως αποτελεί ακόμα αντικείμενο ε, συζήτησης. Αυτό σημαίνει θα είχαμε λιγότερους κανονισμούς, αλλά εγώ πιστεύω ότι για λόγους ορατότητος είναι χρήσιμο να υπάρχουν γενικοί κανονισμοί, οι οποίοι για να βοηθήσουν και την ορατότητα και την απλοποίηση θα καλύπτουν ως το δυνατόν περισσότερα στοιχεία της γενικής λειτουργίας των ταμείων και στη συνέχεια να υπάρχουν επιμέρους ρυθμίσεις για κάθε ταμείο. Εγώ μίλησα με τον Λίκ Φαντερ Μπράντε, τον, τον πρώην πρόεδρο της Επιτροπής των Περιφερειών και του ζήτησα να μου δώσει τις συμβουλές του ώστε να μπορέσει να υπάρξει και μια μεγαλύτερη αντιμετώπιση του θέματος της λεγόμενης πολυεπίπεδης διακυβέρνησης που απασχολεί και την Επιτροπή των Περιφερειών. Για να δούμε σε ποιο βαθμό μπορούμε να ενσωματώσουμε και αυτή την έννοια μέσα στους γενικούς κανονισμούς. Περιμένουμε λοιπόν, να ζητήσαμε να υπάρξει μια πρόταση και από την Επιτροπή των Περιφερειών. Είναι πιθανό βέβαια ότι οι κανονισμοί, ορισμένοι κανονισμοί θα έχουν ουσιαστικά ένα περιεχόμενο δηλωτικού χαρακτήρα και όχι δεσμευτικού χαρακτήρα, αλλά σε άλλες περιπτώσεις νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει και μία, ε, ένας χαρακτήρας πιο δεσμευτικός. Εκεί που χρειάζεται λοιπόν να υπάρχει μία μεγαλύτερη ορατότητα, όταν πρόκειται για τους ε, για τις τοπικές αρχές, τους εκπροσώπους της ε, κοινωνίας των πολιτών κτλ. Είναι απαραίτητο αυτοί να συμμετέχουν στις ε, διαβουλεύσεις για τα μελλοντικά λειτουργικά προγράμματα. Εγώ έχω ακούσει πολλές φορές τις διαμαρτυρίες των περιφερειών ότι το κεντρικό επίπεδο πολλές φορές δεν τους παίζει, δεν τους βάζει στο παιχνίδι. Και από την άλλη μεριά οι κεντρικές κυβερνήσεις λένε πολλές φορές ότι οι περιφέρειες δεν ασχολούνται με τα θέματα αυτά. Επομένως αυτό δεν είναι ένα θέμα το οποίο αφορά μονάχα την ε, Αυστρία και άλλες χώρες τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήταν χρήσιμο να εξασφαλίσουμε τρόπους για να συμμετέχουν όλοι αυτοί οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα θέματα αυτά και κάνω και να κάνω μια έκκληση και προς εσάς ως βουλευτές στις διάφορες επιτροπές τις οποίες είσαστε ενεργοί να μπορείτε να παίζετε το ρόλο των συνομιλητών και να μπορείτε να μας δίνεται ανάδραση σε σχέση με τις ενέργειες και τις προτάσεις της Κομισιόν με στόχο να μπορέσει να υπάρχει αυτή η επαφή με τις ε, τοπικές και περιφερειακές αρχές και να υπάρχει αυτή η λεγόμενη οικειοποίηση ownership της περιφερειακής πολιτικής. Ναι, αλλά εγώ έκανα και μία, διατύπωσα και μία τρίτη ερώτηση, λέει ο κ. Θεωρείτε, κύριε Επίτροπε, ότι ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών μπορεί να είναι σημαντικός, είναι ικανοποιητικός στα πλαίσια της στρατηγικής 2020, ο ρόλος που παίζουν στις κεντρικές στρατηγικές. Αναφέρομαι στο τι συμβαίνει συγκεκριμένα σε τοπικό επίπεδο. Πιστεύω ή μάλλον ελπίζω ότι αυτή η διαδικασία διαπραγματεύσεων θα συμβάλλει στο να υπάρξει καλύτερη ενσωμάτωση και συμμετοχή των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην ε, διαμόρφωση των προγραμμάτων. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την πραγματικότητα λόγω των διαφορετικών παραδόσεων που επικρατούν στα κράτη-μέλη, λόγω της διαφορετικής ε, θέσεις που έχουν οι περιφερειακές και τοπικές αρχές μέσα στη συνταγματική τάξη μιας χώρας και φυσικά και μέσα στη διαδικασία λήψης αποφάσεων. Βλέπουμε ότι υπάρχουν περιφέρειες οι οποίες έχουν πραγματικά σημαντικές πολιτικές αρμοδιότητες σε συνταγματικό επίπεδο και άλλες χώρες όπου ισχύει ακριβώς το αντίθετο. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε πώς θα εξασφαλίσουμε αυτή τη συμμετοχή, γιατί δεν έχουμε ένα ενιαίο χαρακτήρα των, περιφερειακών και τοπικών αρχών. Αλλά ο στόχος μας θα πρέπει να είναι στο βαθμό του δυνατού να μειώσουμε τις ανισομέρειες σε σχέση με το ρόλο των περιφερειακών και τοπικών αρχών, ώστε μέσα σε κάθε κράτος μέλος να μπορέσει να γίνει με τον πιο επωφελή τρόπο αυτή η διαβούλευση. Οι υπηρεσίες μας και οι διαπραγματεύτες μας πάντα θα έχουν σαν στόχο να εξασφαλίσουν την πλήρη συμμετοχή, δεν μπορούν φυσικά να αγγιηθούν ότι αυτά τα πράγματα θα γίνουν από τα κράτη-μέλη με τον επιθυμητό από εμά τρόπο. Θα προσπαθήσουμε όμως και θα το προσπαθήσουμε να το προβλέψουμε στους κανονισμούς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η Κωνσταντσε Κραέλ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Έχουμε συζητήσει για το θέμα αυτό και στο παρελθόν αλλά ήμουνα παρούσα στην τελευταία ε, συνεδρία της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ και ένιωσα ανησυχία γιατί ο Επίτροπος Γεωργίας μίλησε εκεί πέρα για μια καλύτερη μορφή συντονισμού των ε, ενεργειών αγροτικής ανάπτυξης, του Αγροτικού Ταμείου Ανάπτυξης με το Ταμείο Συνοχής. Και θεώρησε ότι πρέπει ορισμένες ενέργειες να χρηματοδοτούνται και από τα δύο ταμεία και από το Ταμείο Συνοχής και από το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Εμείς δεν θέλουμε κάτι τέτοιο. Εμεί θέλουμε να υπάρξει μια μεγαλύτερη επικέντρωση των πόρων του Ταμείου Συνοχής στους αστικούς χώρους και στις άλλες ε, ε, προτεραιότητές μας και να υπάρχει μια καλύτερη συνεργασία με το Αγροτικό Ταμείο για να δημιουργήσουμε περισσότερους χώρους που είναι ανεξάρτητοι. Εσείς δεν έχετε μιλήσει για το θέμα αυτό του συντονισμού με το Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά πώς είναι τα πράγματα στις συζητήσεις που λαμβάνουν χώρα αυτή τη στιγμή στην Κομισιόν και συμμερίζεστε την άποψή μας ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποιο κάποιος ελεύθερος χώρος στον προϋπολογισμό, ώστε το Ταμείο συνεχίζει να μην ασχολείται μόνο με τον αγροτικό χώρο. δεν γνωρίζω μάλλον τις προτάσεις του κυρίου Τσόλος. Ξέρω ότι είναι φανερό ότι έτσι που τις παρουσιάζεται εγώ δεν μπορώ να τις συμμεριστώ. Αλλά στη συζήτηση στην Κομισιόν δεν έχει ακόμα φτάσει σε επίπεδο συζήτησης. Μπορεί να είναι μια πρωτοβουλία απλώς. Εμείς θέλουμε να έχουμε ένα στρατηγικό πλαίσιο στα πλαίσια της Κομισιόν, μέσα στο οποίο η γεωργία, η αλληλεία, η διαρθρωτική πολιτική και το Κοινωνικό Ταμείο που έχουν τέσσερις αρμόδιους επιτρόπους. Οι τέσσερις αυτοί οι επίτροποι που διαχειρίζονται αυτά τα ταμεία έχουν δεσμευτεί να προσπαθήσουμε ενώπιον των άλλων συναδέλφων στην Κομισιόν να παρουσιάσουμε ένα κοινό στρατηγικό πλαίσιο για τον τρόπο με τον οποίο οι διάφορες αυτές μορφές διαρθρωτικών ταμείων θα μπορέσουν να λειτουργήσουν για να υπάρχει μια σαφής στοχοθεσία. Ο στόχος μας προφανώς είναι να αποφύγουμε τις ε, επικαλύψεις και αυτός είναι και ο στόχος των συζητήσεων που λαμβάνουμε χώρα μεταξύ αρμοδίων γενικών διευθύνσεων, γιατί έχουμε πάντα επικριθεί στο παρελθόν ότι μεταξύ του, των αξώνων 3 και 4, δηλαδή του Ταμείου για την Αγροτική Ανάπτυξη και του Ταμείου Συνοχής ή Περιφερειακού Ταμείου υπάρχουν επικαλύψεις. Οι στοχοθεσίες μας λοιπόν θα πρέπει να είναι ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε καλά τα χωράφια μας για να είμαστε καλοί φίλοι και καλοί γείτονες. Να μην υπάρχουν λοιπόν ε, επικαλύψεις, να συζητήσουμε τα πράγματα αυτά με έναν τρόπο ο οποίος είναι επωφελής και όχι να επεμβαίνουν παραπάνω από ένα ταμείο σε ένα και το αυτό πρόγραμμα ή σχέδιο. Αυτή είναι η κατεύθυνση λοιπόν που ακολουθούν οι συζητήσεις στην ε, Κομισιόν. Ελπίζω ότι θα προχωρήσουν αυτά τα πράγματα. Τώρα σας ευχαριστώ βέβαια και την πληροφορία που μου δώσετε ένα πρόσθετο ερώτημα για το στρατηγικό αυτό πλαίσιο. Τι βαθμό δεσμευτικότητας θα έχει και πώς θα σχετίζεται με το γενικό κανονισμό που αναφέρατε. Θα κάνετε ένα περαιτέρω γενικό κανονισμό ή θα συμπεριληφθούν αυτά στον κανονισμό το γενικό που αναφέρατε. Εγώ θέλω να είμαι το η αιχμή του δόρατο στα θέματα της ε, μεταρρύθμισης για τα θέματα αυτά. Δεν ξέρω αν θα μπορέσω να το κάνω και δεν γίνονται αυτά τα πράγματα από τη μια μέρα στην επόμενη. Τι θα επιτύχουμε να έχουμε σε αυτό το γενικό στρατηγικό πλαίσιο. Εμείς ο στόχος μας είναι να ξεκαθαρίσουμε καταρχήν ποιος κάνει τι, ποιες είναι οι αρμοδιότητες του, του κάθε ταμείου και πώς θα λειτουργούν τα πράγματα αυτά στην πράξη και στην εφαρμογή θα, θα το δούμε στην πράξη στο μέλλον. Στην επόμενη δηλαδή χρονική περίοδο προγραμματισμού θα πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω εξελίξεις. Εγώ βλέπω αυτό το οποίο ε, λέτε ότι οι διαφορετικές αυτές στοχοθεσίες δεν είναι απλό να συμπεριληφθούν σε ένα κανονισμό και μόνο. Αλλά ορισμένοι μπορεί να έχουν και διαφορετικές απόψεις για το θέμα αυτό. Από την ομάδα Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε και ευχαριστούμε πολύ τον Επίτροπο που ξαναήρθε εδώ να μας επισκεφθεί και να μιλήσουμε στα πλαίσια της Επιτροπής μας. Πρώτη ερώτηση. Είναι μια ερώτηση που αφορά την ε, δυνατότητα και ικανότητα συνεργασίας. Δηλαδή, ε, τα κονδύλια τα οποία δεν θα έχουν χρησιμοποιηθεί ε, θα μπορούν να επανακατανεμηθούν κυρίως δε να δοθούν ε, στις χώρες οι οποίες καλύτερα έχουν υλοποιήσει τα προγράμματα της στρατηγικής 2020. Ε, επίσης, ποια είναι η άποψή σας ε, για τους δείκτες τους οποίους θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για να διαπιστώσουμε κατά πόσο λειτουργεί η στρατηγική αυτή. Όσον αφορά το πρόγραμμα Interreg, στην περίοδο προγραμματισμού υπήρξαν προβλήματα Τώρα γίνεται μια προσπάθεια να διαπιστώσουμε ποια είναι η καλύτερη προσέγγιση. Η επόμενη, στην επόμενη προγραμματική περίοδο θα πρέπει βεβαίως να ληφθούν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του προγράμματος ε, Interreg. Και η τελευταία μου ερώτηση αφορά το άρθρο 74. Ε, μαθαίνουμε ότι στην τελευταία προγραμματική περίοδο οι ορεινές περιοχές και οι, τα νησιά θα ληφθούν καλύτερα υπόψη. Αλλά δεν μας λέτε και κάτι πιο συγκεκριμένο. Τι ακριβώς θα γίνει. Äh, Για το πρώτο σας ερώτημα. Εξακολουθεί η κατάσταση να είναι τέτοια που η διαδικασία κλεισίματος ουσιαστικά ενός ε, προγράμματος κρατάει και μετά από το τέλος της ε, ε προγραμματικής περίοδου. Υπάρχουν παραγωγικά προγράμματα τα οποία ε, περιλαμβανόντουσαν μέσα στη χρονική περίοδο που τελείωνε το 2006 και η διαδικασία κλεισίματός τους κράτησε και μέχρι σήμερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μπορεί να υπάρξει αυτό το πρόβλημα με τα κονδύλια λόγω του γεγονότος ότι έχει ξεπεραστεί η χρονική περίοδος εφαρμογής ενός προγράμματος. Στο μέλλον φοβάμαι ότι και εκεί θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε περαιτέρω προβλήματα λόγω της ε, στενότητας του προϋπολογισμού. Θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε τέτοια προβλήματα. Όταν όμως δεν έχει υπάρξει πλήρης ε, <clears throat> εξάντληση των κονδυλίων, πολλές φορές το καταλαβαίνουμε αυτό μονάχα στο τέλος ενός προγράμματος και δυστυχώς αυτό δεν μας επιτρέπει να, κατανέμουμε τα κονδύλια. Τώρα μίλησα ιδιαίτερα για το θέμα των δικτών, της ανάγκης να αναπτύξουμε δίκτες οι οποίοι δεν είναι απλώς κάτι το οποίο ε, βρίσκεται πάνω σε ένα φύλλο χαρτί, αλλά είναι πραγματικά ε, γνώμονες καταμέτρησης της επιτυχίας ενός προγράμματος και της επιτυχίας ή όχι ορισμένων διαδικασιών που έχουν να κάνουν με την αύξηση της αποδοτικότητας σε ενεργειακή χρήση κτλ για το πρόγραμμα Interreg που αναφέρατε, τα προγράμματα μάλλον του Interreg. Εγώ φαντάζομαι ότι θα πρέπει να υπάρξει ειδική ρύθμιση για το ε, Interreg που λαμβάνει υπόψη και την αναλογικότητα και πιστεύω ότι σε επόμενους ε, μήνες, στις επόμενες εβδομάδες θα λάβουν χώρα και πιο ενδελεχείς συζητήσεις σε σχέση με τα προγράμματα αυτά του Interreg. Στο τελευταίο σας ερώτημα τώρα. <clears throat> Υπάρχει ήδη και θα υπάρχει και στο μέλλον, έτσι θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον, ένα σύνολο κανόνων για άρεοκατοκιμένες περιοχές. Αυτό αφορά το βόρειο τμήμα της Ευρώπης, τη Σκανδιναβία, όπως σωστά αναφέρατε, ότι αυτό είναι κάτι το οποίο περιέχεται και στη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξασφαλίζεται από την ε, συνθήκη και τα διάφορα ολοκληρωμένα προγράμματα ήδη από το 2008-2009 έχουν προσπαθήσει να αντιμετωπίσουν την προβληματική περιοχών που είναι μειονεκτικές για την νεορινές περιοχές ή νησιωτικές περιοχές. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια συγκεκριμένη χρηματοδότηση γιατί αυτές οι περιοχές περιλαμβάνονται σε ευρύτερες περιφέρειες και εναπόκειται στην αυτονομία των περιφερειών να, των μεγαλύτερων αυτών περιφερειών να κατανείμουν αυτή τη χρηματοδότηση και νομίζω ότι έτσι θα παραμείνει και στο μέλλον. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, ευχαριστούμε που ήρθατε εδώ Έχω αρκετές ερωτήσεις. Ε, πρώτα απ' όλα για τις ε, βιομηχανίες για τις δημιουργικές ε, ε, επιχειρήσεις ε, στα πλαίσια μιας αναπτυξιακής πολιτικής πώς προτίθεστε να τις βοηθήσετε. Επίσης, στα πλαίσια του στόχου 3 βλέπουμε ότι υπάρχουν όλο και περισσότερα προγράμματα, προγράμματα των μεγάλων, των μακροπεριφερειών που βεβαίως θα δημιουργήσουν νέα δραστηριότητα στο τομέα αυτούς. Και η ερώτησή μου λοιπόν είναι διτή για την επόμενη προγραμματική περίοδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σκοπό να δώσει περισσότερους πόρους στον στόχο 3 και επίσης ε, αυτή η έννοια της, ε, ε, της, του, αποθέματος ενέργειας που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, αυτό που αναφέρατε εσείς, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για τον στόχο 3. Äh, Το γενικό θέμα του πολιτιστικού τομέα. Αυτό δεν είναι που θέσατε καταρχήν, αν κατάλαβα καλά. Uh, uh, Το πρώτο σας ερώτημα ήταν για τον πολιτιστικό τομέα. Υπάρχει μία έκθεση πρωτοβουλίας που συζητήσαμε χθες στην Επιτροπή στην Επιτροπή Πολιτισμού ε, βάσει των οποίων υπάρχουν κάποιες ε, επιχειρήσεις οι οποίες δημιουργούν πολιτισμό, ε, δημιουργούν διάφορα πολιτιστικά προϊόντα, ταινίες και άλλα. Κατά την άποψή μας αυτού του είδους η παραγωγή συμμετέχει στην αναπτυξιακή ικανότητα που μπορεί να αναπτύξει μια περιφέρεια. Ε, μια περιοχή και πιστεύουμε ότι αυτό θα πρέπει σαφέστερα να αναφέρεται ε, και να λαμβάνεται υπόψη ενδεχομένως ε, στον περιφερειακό προγραμματισμό. Και αν ρωτώ λοιπόν εάν αυτού του είδους οι επιχειρήσεις και αυτού του είδους η λογική μπαίνει στις επόμενες προγραμματικές περιόδους. Αυτό το θέμα θα πρέπει να αντιμετωπιστεί υπό το πρίσμα της ε, ε, υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Μπορούμε να σκεφτούμε τη δημιουργία ενός συμπλέγματος, ενός κλάστερ για μια συγκεκριμένη περιοχή ή για μια ομάδα περιφερειών και περιοχών. Και εδώ το βασικό ζήτημα είναι να μπορέσουμε να ενισχύσουμε συγκεκριμένες δραστηριότητες, παραδείγματος χάρη παραγωγή ταινιών σε περιοχές οι οποίες έχουν μια ειδίκευση σε τέτοιου είδους καλλιτεχνική και δημιουργική παραγωγή και μπορούν να αποτελέσουν κέντρο για να προσκαλέσουν και άλλες περιοχές να συμμετάσχουν σε αυτή τη ε, διαδικασία με το πλεονέκτημα ότι δεν θα κινδυνεύσει η λειτουργία αυτών των, αυτού του καλλιτεχνικού και πολιτιστικού τομέα στο μέλλον. Υπό το πρίσμα της ειδίκευσης η οποία θα πρέπει να λάβει χώρα στην Ευρώπη μεταξύ των περιφερειών, αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη και η εδαφική συνεργασία που προβλέπεται στον πυλώνα 3 θα πρέπει να αποτελέσει μια πραγματικότητα. έχουμε 2,5% του συνολικού προϋπολογισμού χρηματοδότηση για αυτό το τομέα, περίπου 8 δισεκατομμύρια ευρώ συνολικά. Δεν ε, μπορώ να σας πω ποιος θα είναι ο προϋπολογισμός ο συνολικός της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο μέλλον και επομένως δεν μπορώ να κάνω κάποια συγκεκριμένη δέσμευση για τα θέματα αυτά. Αλλά πιστεύω ότι το ποσοστό αυτό το οποίο το οποίο είναι στη διάθεσή μας για το τομέα αυτό το πολιτιστικό δεν μας επιτρέπει να καλύψουμε οριζόντια προγράμματα που να καλύπτουν όλο το έδαφος της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά τα χρήματα αυτά θα πρέπει κυρίως να βοηθήσουν να υπάρχει καλύτερη συνεργασία αλλά φυσικά έχουμε ήδη ένα μεγάλο αριθμό συμπράξεων και συνεργασιών που ξεκινάει από περιφέρειες που είναι όμορες και εκτείνεται μέχρι τη μακροπεριφερειακή στρατηγική. Πρέπει λοιπόν οι ίδιες οι περιφέρειες να λάβουν υπόψη αυτό το στοιχείο και να χρησιμοποιήσουν μέσα στα λειτουργικά τους προγράμματα ένα τμήμα του προϋπολογισμού τους για να εξασφαλίσουν συνεργασίες οι οποίες είτε υπάρχουν ήδη είτε είναι εν εξελίξη προβλέπονται για το μέλλον. Αυτή είναι και η αντιμετώπιση που έχουμε για τις μακροπεριφέρειες. Δεν πρόκειται για πρόσθετα χρήματα, πρόκειται για χρήματα τα οποία υπάρχουν και τα οποία με μια ευφυά μέθοδο συντονισμού θα πρέπει να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και να χρησιμοποιούνται με πιο επωφελή τρόπο. Έχουμε πολλές λοιπόν περιπτώσεις διαμεθοριακής συνεργασίας στην Ευρώπη και θα πρέπει να καταστεί δυνατό μέσα στη λειτουργική σχεδίαση η κάθε περιφέρεια να λάβει υπόψη αυτό το στοιχείο και να προβλέψει αντίστοιχα κονδύλια μέσα από τη χρηματοδότησή της. you, dear I just... Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να πάρετε σοβαρά αυτό που θα σας πω τώρα. 13 άτομα έχουν εγγραφεί στον κατάλογο. Αν θέλετε να υποβάλλετε ερωτήσεις προς τον Επίτροπο και να σας απαντήσει, θα έχετε στη διάθεσή ένα λεπτό και δύο λεπτά ο Επίτροπος για να την απαντήσει. Διαφορετικά θα παραμείνει ο, ο κατάλογος δίχως να ολοκληρωθούν οι παρεμβάσεις. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα ανάμεσα μας. Τώρα, στο Συμβούλιο και στην Κομισιόν διεξάγεται συζήτηση αναφορικά με το πακέτο που αφορά στις υποδομές. Και εδώ υπάρχει μια νέα προσέγγιση η οποία διαφέρει με αυτήν του παρελθόντος και μιλάμε για νέες ε, ενδεχόμενες χρηματοδοτήσεις. Υπάρχουν ε, πολλοί που είναι υπέρ ενό νέου μέσου το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση αυτού του πακέτου αλλά υπάρχουν και άλλες απόψεις οι οποίες ε, θέλουν να παραμείνει ο υφιστάμενος ε, προϋπολογισμός για τη θέματα συνοχής. Η χώρα μου είναι υπέρ της συνέχισης. Ευχαριστώ. Της μη Και είμαι και Πολωνή. Καλή μπάχα. Äh, Πάρα πολύ σύντομα. Το ερώτημα το οποίο ετέθη σε κάποιο βαθμό προηγουμένως, σε ποιο βαθμό η πολιτική του πολιτιστικού χώρου λαμβάνει υπόψη στη στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Δούναβη, την περιοχή του Δούναβη και αν θα υπάρχουν ειδικοί πόροι για αυτόν τον τομέα. Ο Χέρμαν Βίνκλερ έχει το λόγο, χωρίς μικρόφωνο. Πρώτο ερώτημα. Τα συμπέρασματα τη πέμπτη έκθεση συνοχή τη Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάει για ορισμένε προτεραιότητε για τη μελλοντική ανάπτυξη των περιφερειών και των κρατών μελών. Εγώ θεωρώ ότι είναι πολύ καλό το να υπάρχει κάποια σύνδεση με την Ευρώπη 2020. Αλλά όταν ε, αντιμετωπίζονται το θέμα των προτεραιοτήτων των περιφερειών θα είναι κάτι το οποίο θα το αποφασίσουν οι περιφέρειες, παραγωγικά λαμβάνοντας υπόψη και προβλήματα δημογραφίας κτλ. ή θα επιβάλλονται εκ των άνω. Ένα περαιτέρω θέμα είναι το θέμα της ισοδικίας. Θέλουμε κατά την επόμενη χρονική διάρκεια α, των ε, πρόπτικων να υπάρξει μια διατήρηση των ε, υπεσχημένων. Έχετε μιλήσει και για τα ταμεία καινοτομία. Είναι κάτι το οποίο θα τροποποιηθεί όμως τώρα με την τωρινή αλλαγή των κανονισμών και θα υπάρξει και αναθεώρηση των κονδυλίων που θα αναφέρονται σε αυτούς τους καινοτόμους τομείς. Ähm, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αντιμετωπίσω περισσότερο το θέμα των ακριτικών περιοχών. Ξέρουμε ότι αυτές οι περιοχές είναι γενικά υπολοιπόμενες σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης στην Ανατολική Ευρώπη και θα ήθελα να ξέρω κατά πόσον εσείς θέλετε να ακολουθήσετε μια συγκεκριμένη πολιτική σε σχέση με αυτές τις περιοχές μέσα στα, στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής και ποια θα είναι η αντιμετώπιση σας, ποια είναι η αντιμετώπιση που θέλει να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να υποστηρίξει αυτές τις ασθενείς περιοχές. Στην κυρία Κολάσκα Μπομπίνσκα, η οποία ίσως ε, κάποιος θα της μεταφέρει την απάντηση. Υπάρχουν πράγματι πολλές συζητήσεις για το πώς θα μπορέσουμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες, ιδίως για θέματα υποδομών. Πράγματι, συζητάτε και το θέμα των project bonds, των ε, ευρωομολόγων για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων σχεδίων που θα εξασφαλίσουν ένα συγκεκριμένο εισόδημα. Εγώ δεν έχω τίποτα εναντίον του να υπάρξει μια τέτοια ρύθμιση αν έχει προετοιμαστεί αυτό το εγχείρημα με σωστό και θετικό τρόπο. Αυτό θα ενισχύσει τις προσπάθειές μας, πιστεύω. Δεν πρόκειται μονάχα για το θέμα της χρηματοδότησης, αλλά και της διαμόρφωσης των προγραμμάτων αυτών, ώστε να είναι ε, εφαρμόσιμα. Γιατί το είπα και προηγουμένως, πολλές φορές τα προγράμματα δεν αποτυγχάνουν λόγω έλλειψη χρημάτων, αλλά λόγω άλλων παραγόντων. Στα θέματα λοιπόν των μεταφορών, εγώ συμφωνώ με τον κύριο Κάλλας ότι θα πρέπει να έχουμε αυτή την κοινή στρατηγική προσέγγιση σε σχέση με τα υποδείγματα που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε για την ε, μεταφορά παραδείγματος από τις οδικές μεταφορές, τις σιδηροδρομικές μεταφορές, την κατασκευή των αντιστοίχων υποδομών, ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις περιφέρειες με μια κοινή αντιμετώπιση και όχι να περιοριστούμε μονάχα στα προγράμματα τα 10 αλλά να δούμε και πώς επηρεάζουν αυτά τα σχέδια της ε, περιφέρειας. Και το ίδιο ισχύει και για θέματα όπως αυτά της τροφοδοσίας ε, με ενέργεια. Θα πρέπει και εδώ να αναπτύξουμε νέα πρόσθετα υποδείγματα χρηματοδότησης. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Ο στόχος μας είναι να συνδέσουμε όλες, αυτά, όλες αυτές τις ψηφίδες με ένα τρόπο αποτελεσματικό. Για τα θέματα πολιτισμού έχω ήδη μιλήσει. Ξέρω ότι η στρατηγική του, της περιοχής του Δούναβη περιλαμβάνει κάποιες ε, δραστηριότητες αυτού του είδους. Τώρα δεν ξέρουμε ακόμα για τη χρηματοδότηση, θα πρέπει να είναι το αντικείμενο συμφωνίας, αλλά υπάρχουν πολλά προγράμματα τα οποία έχουν υποβληθεί. Πιστεύω ότι θα πρέπει να είναι δυνατόν να γίνει μια τέτοια χρηματοδότηση του πολιτιστικού τομέα. Αυτό είναι θέμα ευφυ ευφυούς ε, χρηματο... των κονδυλίων. Το ερώτημά σας ε, κύριε Βίντλε, μιλήσατε για την τροποποίηση ορισμένων κανόνων για τα προγράμματα του, στο περιφερειακό επίπεδο. Υπάρχουν πολλά από αυτά τα προγράμματα τα οποία εντάσσονται στην στρατηγική της Ευρώπης 2020. Ο στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε ότι από τη μία πλευρά θα έχουμε μια καλύτερη ορατότητα των αποτελεσμάτων και από την άλλη πλευρά θα υπάρχει καλύτερη ορατότητα από την πλευρά των πολιτών για τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται τα χρήματα του, του Ταμείου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και επομένως είναι οι περιφέρειες οι οποίες θα πρέπει να αποφασίσουν επί τη βάση των αναγκών τους πώς θα χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια και ποιε θα είναι οι προτεραιότητε. Από τη δική μας πλευρά, βέβαια, εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα βελτιώνεται η ποιότητα των ε, προγραμμάτων αυτών. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να έχουμε τη δυνατότητα μετά από ένα χρονικό διάστημα, 7 χρόνια παραδείγματος χάρη, να καταμετρήσουμε την πρόοδο η οποία έχει επιτευχθεί και να ξέρουμε αν θα πρέπει να τροποποιήσουμε την κατεύθυνση της χρηματοδότησης, αλλά το ουσιαστικό είναι να μπορούν οι περιφέρειες να γνωρίζουν ποιες θα είναι οι προτεραιότητές τους. Όπως είπατε βέβαια χρειάζεται μια σταθερότητα. Δεν ε, έχω διαφορετική άποψη, αλλά αυτός είναι ένας τομέας στον οποίο έχουμε ήδη αποκομίσει ορισμένα διδάγματα Πολλές φορές στο παρελθόν υπήρξε η ανάγκη να αντλήσουμε συμπεράσματα και να τροποποιήσουμε τις διαδικασίες μας και τις κατευθύνσεις μας μέσα σε μια περίοδο προγραμματισμού και όχι να περιμένουμε μέχρι το τέλος της δημοσιονομικής περίοδου. Η αντιμετώπιση της Επιτροπής μου είναι ότι πρέπει να υπάρχει μια αντιμετώπιση στην, στο λεγόμενο shared management, να υπάρχει μια κοινή αντιμετώπιση σε ό,τι αφορά χάρη τη χρήση ενδιαμέσων φορέων χρηματοδότησης. Ο στόχος μας όμως είναι να διαμορφώσουμε ευρωπαϊκά πρότυπα ενιαία μέσα στα οποία μπορούν να υπάρχουν ε, εξαιρέσει αν αυτό είναι απαραίτητο, αλλά να κινούμαστε για, μέσα στα πλαίσια αυτά. Για τις ε, ακριτικές περιοχές, όπως γνωρίζετε, υπάρχουν πολύ διαφορετικά προγράμματα τα οποία αντιμετώπισαν ακριβώς δυσκολίες εφαρμογής λόγω της πολυπικιλίας των περιοχών αυτών που είναι οι ακριτικές περιοχές, οι εξωτερικές περιοχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αλλά εμείς προσπαθούμε όσο το δυνατόν να βγούμε από αυτές τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε στο παρελθόν ώστε να υπάρξει μια σωστή εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων και να συνεργάζονται αυτές οι, οι ιδιαίτερες περιοχές με παραμεθόριες περιοχές οι οποίες είναι εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μέσα στα γεωπολιτικά συμφέροντα τη Ευρωπαϊκή ένωση να προωθήσουμε τέτοιου είδου σχέσει και συνεργασίες. Η κυρία Ένστα. Εγώ σας ευχαριστώ για την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας. Δεν γίνεται σε κάθε επιτροπή μια τόσο ενδελεχή συζήτηση. Έχω δύο ερωτήματα. Το πρώτο ερώτημα. Το πρώτο αφορά λοιπόν το σύνολο του, της προβληματικής γιατί η συγχρηματοδότηση είναι σαφέ ότι πρέπει να παραμείνει η συγχρηματοδότηση. Είναι σημαντικό στοιχείο για το μέλλον. Εσείς λέτε ότι θα πρέπει να υπάρξει και το ποσοστό συγχρηματοδότησης αντικείμενο επανεξέτασης. Θα ήθελα να ξέρω ακριβώς τι προβλέπετε να κάνετε στον τομέα αυτό των ποσοστών συγχρηματοδότησης. Το δεύτερο θέμα το οποίο θα ήθελα να θίξω Αναφερθήκατε στη χρήση καινοτόμων εργαλείων χρηματοδότησης. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον για μένα. Στην Γερμανία ξέρω ότι υπήρξαν παραδείγματα επιτυχούς χρήσης τέτοιων εργαλείων. Το ερώτημα για μένα πώς προβλέπετε να γίνει αυτή η χρησιμοποίηση και επίσης αν αυτό θα σημαίνει ότι αυξάνεται το πεδίο εφαρμογής αυτών των ε, εργαλείων. Μήπως μπορείτε να μου εξηγήσετε καλύτερα ποια είναι η πρόβλεψή σας σε σχέση με αυτά τα καινοτόμα εργαλεία. Η Ελίζα Μπεσουσέτερ. Καλημέρα κύριε Επίτροπε. Σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Και θέλω να σας ευχαριστήσω επίσης για την πολύ καλή παρουσίαση που μας έχετε κάνει των θέσεων της Κομισιόν για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η περιφερειακή πολιτική στο μέλλον και σας συγχαίρω για την ανακοίνωση αυτή που κάνατε χθε, γιατί σα ήταν ο πρώτο επίτροπο μετά από 15 χρόνια που κάνετε το θάρρο να κάνετε μία δήλωση για την πολιτική συνοχή και την αηφορία τη. Τώρα το ερώτημα είναι, αυτά τα οποία είπατε στην ανακοίνωσή σας θα αντανακλώνται στον γενικό κανονισμό και θα είναι πραγματικά υποχρεωτικές ε, ρήτρες για τα κράτη-μέλη και τι προβλέπεται για το λεγόμενο απόθεμα αποδοτικότητας, δηλαδή το πρόσθετο αυτό μπόνους το οποίο μπορεί να δώσει η Κομισιόν. Εγώ πιστεύω ότι αυτό είναι ένα από τα καλύτερα εργαλεία που μπορεί να έχετε στη διάθεσή σας ως Κομισιόν για να εξασφαλίσετε την ποιότητα των προγραμμάτων αυτό το ε, επίδομα αποδόσης Έχω δύο ερωτήσεις, Πρόεδρε. Η μία είναι περισσότερο πολιτικό χαρακτήρα. Τελείωσε η τάση να τίθεται η πολιτική συνοχή σε συνδυασμό με την ε, στρατηγική του 2020 που αφορά τον ε, ανάπτυξη το Φόρουμ Συνοχής ε, νομίζω ότι ασχολείται με τρία ζητήματα, δηλαδή i αηφόρου και ανταγωνιστικότητα. Αυτή η τάση λοιπόν έχει τελειώσει, έχει ολοκληρωθεί, διότι νομίζω ότι η τάση αυτή ήταν ε, εσφαλμένη τώρα. Κάτι για την ατζέντα. Ακούσαμε τον αριθμό των κανονισμών, αλλά ποια είναι η πρόθεσή σας. Ε, νομίζω ότι θα είναι καλύτερη στιγμή να θέσετε επιτάπητος ε, τους κανονισμούς ε, και στο πλαίσιο του συζήτηματος με το Κοινοβούλιο. Θα, πρέπει στην αρχή να υπάρξει η δημοσιονομική πρόβλεψη από την Κομισιόν και μετά να περάσουμε στην εξέλιξη των κανονισμών. Ή θα πρέπει να προχωρήσουν παράλληλα. Χθε το απόγευμα έθεσα κάποιε ερωτήσει στον Ούγκρο Πρόεδρο. Αποφάσει που αφορούν την περίοδο των ε, προβλέψεων. έχουμε πενταετή περίοδο, τότε η πολιτική, το σύνολο της πολιτικής θα πρέπει να τροποποιηθεί. Λοιπόν, πρόκειται για μια απόφαση η οποία δεν έχει ληφθεί ακόμα και η ερώτησή μου είναι εξή. Τι γίνεται με την ατζέντα και αν νομίζετε ότι η πρόταση που κάνετε είναι, αποτελεί την βέλτιστη λύση. Ευχαριστώ, Μικαλ Τόιλ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, το ερώτημά μου ακολουθεί την διακατεύθυνση με τον προλαλήσαντα. Μιλήσαμε προηγουμένως για τον προσδιορισμό των κονδυλίων, τώρα μιλάμε για αιρεσιμότητα. Εγώ θα θεωρούσα λανθασμένο η περιφερειακή πολιτική να περιλαμβάνεται μονάχα στο στόχο περιεκτική ανάπτυξη. Εγώ πιστεύω ότι και η ευφυής και η αηφόρος ανάπτυξη είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιτευχθεί στις περιφέρειες και γι' αυτό θα με ενδιαφέρει πάρα πολύ να ξέρω ποια είναι η δική σας άποψη συγκεκριμένα για το εξής ερώτημα βλέπετε τη δυνατότητα μέσα από το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης <clears throat> έχουμε την ανάγκη προσαρμογής στην παγκοσμιοποίηση. Αλλά αν προχωρήσουμε με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε και ένα ταμείο για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, ένα ταμείο προσαρμογή στη δημογραφία κτλ. κτλ. Λοιπόν, δεν θέλω να υπάρξει ένας τέτοιος πολλαπλασιασμός. Έχουμε να αντιμετωπίσουμε τη ρευστότητα του κόσμου σε παγκόσμιες συνθήκες, κλιματικές, τεχνολογικές κλπ. Μήπως όλα αυτά θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε μια συγκεκριμένη και συνολική περιφερειακή και εδαφική αντιμετώπιση. Πώς το βλέπετε αυτό, κύριος Ντεάντζελης. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, εντάχει. Τρία ζητήματα. Πρώτον, για να προωθήσουμε τις ε, παραγωγικές επενδύσεις που κατά μου πρόκειται για επενδύσεις που αφορούν στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Θεωρώ ότι θα πρέπει να εξεύρουμε λίγες προτεραιότητες. Η πρώτη ερώτησή μου λέει εξής. Ποια τι προτεραιότητες και ποια κριτήρια θα εφαρμοστούν προκειμένου να δοθούν ε, ε, να επιβληθούν κυρώσει αλλά και κίνητρα και κάτι ακόμα. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί κανονισμοί, υπερβολικά πολλοί κανονισμοί. Τι μέτρα λοιπόν προβλέπετε για να απλουστεύσετε και να επιταχυνθούν ως εκ τούτου οι διαδικασίες ε, για, την, για τις δαπάνες. Και τρίτη ερώτηση, τι μέσα προβλέπετε για ένα καλύτερο συντονισμό στη χρήση των διαθροτικών ταμείων. Ευχαριστώ. για το ζήτημα της χρηματοδότησης. Θα θυμόσαστε ότι για τις περιοχές της σύγκλησης, της περιφέρειας σύγκλησης, είχαμε προβλέψει αρχικά συγχρηματοδότηση 25% και περάσαμε μετά στο 15%. Και ένα άλλο ερώτημα αφορούσε τις περιοχές του phasing in και του phasing out οι οποίες θα είχαν συγχρηματοδότηση μεταξύ 50% και 75% με την ε, έννοια της ε, περιοχής η οποία υπόκειται σε μεταβατικό, βρίσκεται σε μεταβατικό στάδιο. Εμείς δεν θεωρώ ότι για τις περιοχές αυτές θα πρέπει να μειώσουμε τη συγχρηματοδότηση κάτω από το 50% γιατί είναι απαραίτητο να δώσουμε το σωστό μήνυμα ότι τουλάχιστον το ίμιση ενός σχεδίου ή ενός προγράμματος σε περιφερειακό επίπεδο θα πρέπει να καλύπτεται από τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ μπορώ να κατανοήσω ότι με τη δημιουργία κινήτρων και μπόνους για ορισμένες ε, για ορισμένα εργαλεία και ορισμένα προγράμματα μπορούμε να προβλέψουμε ένα χαμηλότερο ποσοστό συγχρηματοδότησης. Αλλά αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει ακόμα να τα αντιμετωπίσουμε σε πληρέστερη συζήτηση. Εγώ θεωρώ ότι η γενική αρχιτεκτονική του συστήματος είναι σωστή. Μπορούμε να χρειαστεί να κάνουμε κάποιες μικρές αλλαγές. Αυτό το οποίο προβλέπεται αυτή τη στιγμή στον προϋπολογισμό είναι ένα περίπου 3% δηλαδή 10 δισεκατομμύρια και είναι πολύ πιθανό ότι μέχρι το τέλος της περίοδου προγραμματισμού θα έχει εξαντληθεί αυτό το ποσό. Και εμείς θα θέλαμε να αυξηθεί μέχρι και το τετραπλάσιο αυτό το ποσό. Βέβαια, θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Δεν μπορούν όλα τα προγράμματα μέσα στην περιφερειακή πολιτική να προσαρμόζονται σε ένα τέτοιο στόχο. Εξακολουθεί το στοιχείο της χορήγησης πολλές φορές να κυριαρχεί σε ορισμένα είδη προγραμμάτων. Μα ενδιαφέρει, παραγωγός χάρη, θέματα που έχουν να κάνουν με υποδομές παιδείας, με την κατάρτιση στα πανεπιστήμια και σε αυτά δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, τα ανανεούμενα ταμεία, τα revolving funds για την ε, εκπαίδευση. Στις περιπτώσεις λοιπόν αυτές χρειαζόμαστε και στο μέλλον να διατηρήσουμε τις ε, διατάξεις οι οποίες ίσχυαν στο παρελθόν. Μπορούμε να φανταστούμε περαιτέρω καινοτόμε ιδέες, αλλά σε πολλούς τομείς όπως είναι η χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μπορούμε να φανταστούμε καινοτόμε ιδέες. Ο στόχος μας είναι να μπορεί να υπάρξει μια καλύτερη χρηματοδότηση και ένα καλύτερο αποτέλεσμα, αλλά φυσικά αυτό δεν είναι εφικτό σε όλες τις περιπτώσεις για το θέμα της αηφορίας. Σας ευχαριστώ για το πολύ θετικό τρόπο με τον οποίο έχετε αντιδράσει στην πρότασή μας. Πολλές φορές έχουμε δυσκολίες να εφαρμόσουμε αυτές τις έννοιες στην πράξη. Έχουμε προτεραιότητες οι οποίες ουσιαστικά <clears throat> είναι οριζόντιες και διατρέχουν όλες τις προσπαθίες μας όπως είναι η αηφορία. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να βρίσκεται σε όλους τους κανονισμούς μας και είναι τμήμα της εντολής διαπραγμάτευσης που έχει η Κομισιόν στις διαπραγματεύσεις με τις περιφέρειες και τα κράτη-μέλη. Και στον τομέα αυτό έχουμε ένα διψήφιο ποσό το οποίο προβλέπεται για τη χρηματοδότηση των ε, προγραμμάτων. Και φυσικά είναι μια αρχή η οποία υποχρεωτικά θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. <clears throat> το αποθεματικό απόδοσης μπορεί να <clears throat> παίξει κάποιο ρόλο εδώ και ξέρω ότι και το λέω ενώπιον ενό κοινοβουλίου, ξέρω ότι εκεί είναι που αντιμετωπίζουμε πολλές φορές την μεγαλύτερη αντιμετώπιση, αντίδραση από τα κράτη-μέλη. Γιατί τα κράτη-μέλη λένε ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να τα διανύμουν τα κράτη-μέλη τα ίδια. Και έχουν αντίδραση στο να υπάρχει μια απόδοση αυτών των πριμ ουσιαστικά, των πριμ απόδοσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι ένα από τα σημεία τα οποία θα δημιουργήσουν τις μεγαλύτερες διαμάχες ίσως. Και εάν έχω την υποστήριξη του Κοινοβουλίου, νομίζω ότι τα πράγματα θα είναι πολύ πιο εύκολα για μας. Αλλά και εγώ γνωρίζω πολύ καλά ότι είναι μεγάλες οι αντιδράσεις των κρατών μελών και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται παράξενο. Για το θέμα της περιεκτικής ε, ανάπτυξης. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα στο θέμα αυτό, αλλά το επεξεργαζόμαστε και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στο φόρουμ συνοχής και ποιες θα είναι οι βασικές έννοιες οι οποίες θα προέλθουν από το φόρουμ συνοχής. Αν θέλουμε να εφαρμόσουμε αυτή την έννοια <clears throat> της ε, περιεκτικότητος, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να δούμε μια περιοχή μονάχα υπό ένα οπτικό πρίσμα, θα πρέπει να δούμε την ε, συνολική αντιμετώπιση. Θέλουμε λοιπόν μια ολιστική αντιμετώπιση η οποία θα είναι και ευφυής και περιεκτική. Και ξέρω ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι υποσυζήτηση στην Επιτροπή ΣΟΥΡΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτή η γνωμοδότηση της Επιτροπής ΣΟΥΡΕ θα ληφθεί υπόψη. Η δική μας αντιμετώπιση είναι ότι μερικές εβδομάδες μετά την πρόταση για το χρηματοδοτικό πλαίσιο θα έρθουν οι προτάσεις μας για τους κανονισμούς. Πρόκειται να είναι κάποια στιγμή προς τον Ιούλιο, εάν έχουν παρουσιαστεί οι προτάσεις για τα χρηματοδοτικά τον Ιούνιο. Για το σύνολο της, για το χρονικό χρονική διάρκεια της περίοδου, εγώ δεν ξέρω αν θα είναι 5 συν 5 ή κάτι άλλο. Τα 7 χρόνια για μένα είναι το ελάχιστο για μια αποτελεσματική πολιτική. Ίσως θα είναι πιο απλά τα πράγματα αν έχουμε 7 χρόνια και όχι 5 συν 5. Αυτό είναι μια μεγάλη συζήτηση η οποία πρέπει να λάβει η χώρα. Προς το παρόν όμως δεν μπορώ να σας πω τίποτα περισσότερο. Μπορώ να σας πω ποια είναι η δική μου θέση που έχω παρουσιάσει σε διάφορες περιπτώσεις για τα 7 χρόνια. Για, για το επόμενο ερώτημα Αν θέλουμε να έχουμε και άλλα ταμεία, αν θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε τον αριθμό των ταμείων στο ερώτημα του κύριου Τόιρετ, ξέρω ότι πρέπει να διατηρήσουμε ένα επίπεδο ευελιξίας και υπάρχει συζήτηση πάντα στα πλαίσια της Κομισιόν. Δεν έχει ε, έχει νόημα προφανώς από τη μία πλευρά να εξασφαλίσουμε τη σταθερότητα. Γι' αυτό μιλάμε για 7 χρόνια, για μια επαρκή περίοδο προγραμματισμού. Συγχρόνως όμως πρέπει να διατηρήσουμε την απόλυτη ευελιξία, να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε γεγονότα τα οποία συμβαίνουν σε διεθνές επίπεδο και τα οποία απαιτούν από εμά μια ευελιξία στον τομέα του προϋπολογισμού. Δεν μπορούμε να τα προβλέψουμε όλα, δεν μπορούμε να τα έχουμε όλα καλυμμένα αλλά ε, προφανώς εγώ έχω κάνει μια προσπάθεια να σκεφτώ περισσότερο για το πώς θα μπορέσει να λειτουργήσει στο μέλλον και να ε, παίξει κάποιο ρόλο το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση. Ο κύριος Άντορ, ο οποίος είναι αρμόδιος για το Κοινωνικό Ταμείο, είναι και αυτός ο οποίος είναι πιο αρμόδιος για να δει τι προβλέπεται για τις οικονομικές ε, παραμέτρους για την αγορά εργασίας και με το ποιο τρόπο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί πιο επωφελώς το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης. Ευχαριστώ. Η Σοφή Οκόνη έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, σε ευχαριστώ που βρίσκεστε σήμερα ανάμεσά μας για αυτήν την ανταλλαγή απόψεων εντάχει. Θα ήθελα να αναφερθώ για την ε, Νίπεθ, στην Ήπεθρο. Αλλά ωστόσο, θα ήθελα να πω ότι ο όρος Ήπεθρος δεν έχει συμπεριληφθεί στην πέμπτη έκθεση. Θα το θέξουμε μια άλλη φορά το ζήτημα. Σήμερα το πρωί θα ήθελα να μας ε, διαφωτίσετε σχετικά με την άποψή σας αναφορικά με την ενδιάμεση κατηγορία. Πρόκειται για ένα ζήτημα το οποίο ε, απασχολεί ιδιαίτερα πολλές πολιτικές ομάδες και θα ήθελα να μας πείτε πώς βλέπετε τα πράγματα. Αυτή η διάμεση κατηγορία δεν έχει ως στόχο να αφαιρέσει χρήματα από έναν στόχο και να καλύψει κάποιον άλλον αυτόν τον ενδιάμεσο και κατά πόσο είναι συνεκτικό και πιο ασφαλές σε όλη φορά την μακροπρόθεσμη πολιτική συνοχής και την περαιτέρω ενίσχυσή της, αλλά και με μια πολιτική με μεγαλύτερη συνοχή και αλληλεγγύη. Εξηγήστε μας λοιπόν λίγο σχετικά με τον διάμεσο στόχο. Θα ήθελα τώρα να μου απαντήσετε και σε κάτι άλλο αναφορικά με το έρασμος των τοπικών αρχών. Των... Ναι, μπορείτε να συνεχίσετε, όχι δεν θα συνεχίσετε. Το έρασμος των τοπικών ε, αρχόντων είναι ένα ζήτημα απαραίτητο για να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό πνεύμα στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής συνοχής και που θα επιτρέψει να λιάνει κάποιες ε, διαφορές. Ε, είχα ως άποψη να την προωθήσω μέσω του προγράμματος Συντερέλ για να κάνω μια δοκιμή, αλλά είδα ότι τα 2 εκατομμύρια ευρώ που βλέπονταν στον... για τον προπολογισμό δεν υπήρχαν πλέον Μπορούμε λοιπόν να συνεχίσουμε με, αυτή το, αυτόν τον τρόπο. Κοίτα, έψαξα μαζί με τον κύριο Λαμασούρ, δεν τα βρήκαμε αυτά τα 2 εκατομμύρια. Μπορεί να κάναμε και λάθο. Πείτε μα αν θα συνεχίσουμε ή δεν θα συνεχίσουμε αυτή την ε, πολιτική για του ε, τοπικού άρχοντε. Νομίζω ότι είναι πολύ καλό για την πολιτική συνοχή, για την συνεκτικότητά τη απέναντι στους ε, ερετούς άρχοντες οι οποίοι θα πρέπει να ε, συμμετάσχουν σε αυτήν την Ενωμένη Ευρώπη. Ευχαριστώ. Έχουμε ακόμα έξι άτομα. Η Οκίμη παρακαλώ, είστε σύντομος. Ένα ερώτημα μονάχα κυρία Πρόεδρε, αξιότιμε κύριε Επίτροπε. Η Κομισιόν 18 Ιανουαρίου είπε ότι θέλει να αναπτύξει την ευρωπαϊκή διάσταση του αθλητισμού και να προωθήσει την απασχόληση στον τομέα αυτό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και λέει ότι θέλει να χρησιμοποιήσει το Περιφερειακό Ταμείο για την υποστήριξη υποδομών στον αθλητισμό ως εργαλείο για μια περαιτέρω ανάπτυξη στον Περιφερειακό Ταμείο και με τον τρόπο αυτό να ενισχύσει τις δράσεις του Κοινωνικού Ταμείου και τις ικανότητες και δεξιότητες της εργατικής δύναμης που ασχολείται στον τομέα του αθλητισμού. Τα χαιρετίζω όλα αυτά, αλλά τα σχέδια δράση των Δήμων, πολλές φορές και των κοινοτήτων, έχουν μία διάρκεια πέντε ετών. Θα μπορέσουν να ληφθούν αυτά υπόψη για τις υποδομές αθλητισμού από το 2014 για να υπάρξει πρόσθετη χρηματοδότηση των ε, Τη ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν μπείτε ναι σε αυτό το πράγμα θα σα είμαι ιδιαίτερα Ο Λουίς Άλβες. Ε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Εγώ θα έλεγα πάντα ότι έχουμε τέσσερι βασικού στόχου: να λύσουμε το πρόβλημα των δημοσίων οικονομικών, να εξασφαλίσουμε λιτότητα στον προπολογισμό, να δώσουμε δυναμική στην οικονομία και στην απασχόληση και να μειώσουμε τι διαρθρωτικέ ανισομέρειε και τις ανταγωνιστικές ασυμμετρίες και να παίξουμε κάποιο ρόλο στο διεθνή χώρο. Μήπω σα φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε την πολιτική συνοχή για να αντιμετωπίσουμε όλου αυτού του στόχου, ιδίω για τη μείωση των περιφερειακών ασυμμετριών και τη ασυμμετρία στην ανταγωνιστικότητα και στην απασχόληση. Πώ θα μπορούσε λοιπόν να είναι ένα εργαλείο το Ταμείο Συνοχή για να αντιμετωπίσουμε και την κρίση των δημοσίων οικονομικών και να εξασφαλίσουμε τη λιτότητα του προπολογισμού. Αυτό μου φαίνεται κάτι το οποίο είναι αμφισβητήσιμο. Από την άποψη αυτή, ποια είναι η θέση σα σε σχέση με τη χρήση τη αιρεσιμότητα, ιδίω με έναν τρόπο που θα είναι αυτόματο, στα διαρθρωτικά ταμεία, όταν πολλέ φορέ οι περιοχέ αυτέ έχουν πολύ λίγη υπευθυνότητα για τη δημιουργούμενη ανισομέτρια που είναι αντικείμενο των κρατών μελών και όταν δεν έχουν πραγματικό έλεγχο στη χρηματοοικονομική ή οικονομική του κατάσταση και ουσιαστικά εξαρτώνται από τα κράτη-μέλη. Μήπω είναι υπερβολικό αυτό και οδηγεί σε καταστάσει οι οποίε μπορούν να οδηγήσουν σε αδικία. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Σάνσε Σμιτ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για αυτόν τον ε, αποτελεσματικό και καρποφόρο διάλογο. Θα ήθελα να υποστηρίξω αυτό το θέμα των ενδιάμεσων περιφερειών. Θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα των μακροπεριφερειών και να μάθω ποια είναι η προσέγγισή σας πάνω σε αυτό το θέμα που δημιουργεί πολύ χα, ε, χαλαρές αντιδράσεις από πλευράς μας. Πώς βλέπετε λοιπόν αυτήν την, ε, τις στο πλαίσιο της ε, εδαφικής πολιτικής και συνεργασίας. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Να επιτρέψω να μιλήσω ρουμανικά. Θα ήθελα να θέσω μια ερώτηση τεχνικής φύσης. Η Κομισιόν και εσείς ω εκ τούτου ε, προσπαθείτε να βελτιώσετε την κατάσταση των ε, των υπεργολάβων και υπεργολαβιών, διότι το ζήτημα είναι πολύ σημαντικό. Πάρα από ένας πολύ υψηλό ε, αριθμός ε, υπεργολάβων ε, σημαίνει καθυστέρηση αλλά και μεγαλύτερη έξοδα, παράλληλα όμως και διαφθορά, χρηματισμό και πελατειακές σχέσεις. Υπάρχει λοιπόν η δημιουργία μιας πολιτικής πελατειακής πελατείας θα έλεγα. ένα χιλιόμετρο αυτοκινητοδρόμου κοστίζει 83 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο. Κοστίζει λοιπόν 83 εκατομμύρια ευρώ. Είναι δυνατόν. Πρόκειται για ένα παγκόσμιο ρεκόρ. Τι προτίθεστε να κάνετε προκειμένου τα ευρωπαϊκά χρήματα να χρησιμοποιούνται με τρόπο πιο έντιμο. The last question from Derek Vaughan. Derek Vaughan, τελευταία ερώτηση. Ευχαριστώ. Θα είμαι πολύ σύντομος. Ο Επίτροπος ε, πέτυχε πολλά μέχρι τώρα και θα ήθελα να τον συγχαρώ για όλα όσα πέτυχε. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις όμως που φορούν λεπτομέρειες και μία από αυτές ε, αφορά το ζήτημα των αστικών περιφερειών. Οι αστικές περιοχές θεωρούνται ως ε, μια οικονομική δύναμη αλλά θα ήθελα να μας δώσετε έναν ορισμό σχετικά με τις περιοχές αυτές. Αυτός είναι ένας τομέας όπου τα κράτη-μέλη και οι περιφέρειες θα πρέπει να δείξουν μια ευελιξία προκειμένου να προσδιορίσουν αυτές τις αστικές περιοχές. Äh, äh, Ευχαριστώ. Να απαντήσω στον κύριο Ντεάντζελης πρώτα. λέτε ότι έχουμε τόσο πολλούς κανονισμούς που αυτό δημιουργεί πρόβλημα. Στην τελευταία προγραμματική περίοδο σε ό,τι αφορά την περιφερειακή πολιτική, η κυρία Χίμπνερ έκανε μια υποδηματική προσπάθεια να περιοριστεί ο αριθμός των προγραμμάτων στην πολιτική συνοχής και στην πολιτική περιφερειακών θεμάτων. Αυτό είναι ένα παράδειγμα το οποίο μπορείτε να λάβετε υπόψη. Ο καθένας φυσικά πρέπει να συμβάλλει σε αυτή την προσπάθεια. Σε ό,τι αφορά το, τη χάραξη των προτεραιοτήτων, θέλω να επαναλάβω αυτό που είπα προηγουμένως, θα πρέπει να είναι λίγες οι προτεραιότητες στις περιοχές του στόχου ανταγωνισμού με σαφή ε, στοχοθεσία θα πρέπει οι περιοχές αυτές να επιλέξουν ποιοι είναι οι στόχοι που θέλουν να εξασφαλίσουν. Να υπάρχει λοιπόν ένα μενού από το οποίο να μπορέσει να γίνει μια επιλογή, αλλά στη συνέχεια οι περιοχές είναι αυτές οι οποίες θα πρέπει να προτείνουν. για τους κανονισμούς. Υπάρχει πάντα αυτή η κριτική ότι προσπαθούν να ρυθμίσουν τα πάντα. Είναι ε, ορατό αυτό ότι πάρα πολλοί θεωρούν ότι είναι υπερβολικά αυτά τα οποία θέλουν να ρυθμίσουν οι κανονισμοί. Αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχουν τα παραθυράκια τα οποία δημιουργούνται αν κάποιος δεν ρυθμίζει τα πάντα και μας υποχρεώνουν να λάβουμε υπόψη την ανάγκη να μην υπάρχουν τέτοια παραθυράκια. Επομένω, είναι χρήσιμο να δούμε του κανονισμού και να δούμε τι μπορούμε να διαγράψουμε από τι λεπτομέρειε. Από την άλλη πλευρά, δεν θέλουμε να αφήσουμε πράγματα τα οποία μένουν ε, χωρίς κάποια ρύθμιση και τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν με τρόπους που δεν μπορούμε να του προβλέψουμε εκ των προτέρων. Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα λοιπόν στην πολιτική περιφερειακών θεμάτων να εξισορροπήσει τις δύο αυτές μέρημνες και να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε κοινά ευρωπαϊκά πρότυπα. Και το έχω πει αυτό και στην Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού και έχω ζητήσει και την υποστήριξη τη δική σας και την η επίλυση των προβλημάτων δεν μπορεί να προέρχεται από αυτοσχέδιες λύσεις. Εμείς θα πρέπει να προσπαθούμε να λύσουμε όλα αυτά τα προβλήματα. Είναι ίσως μια εργόδης και δύσκολη διαδικασία, αλλά αυτό είναι απαραίτητο για να έχουμε μια σωστή αντιμετώπιση. Υπάρχουν προβλήματα και επιτοπίως, υπάρχουν και προβλήματα στις Βρυξέλλες. Ο στόχος μας λοιπόν είναι να δούμε πώ θα αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο τρόπο από τη δική μας πλευρά το κάθε πρόβλημα. Οι ενδιάμεσες κατηγορίε τώρα, όπως αναφέρεται το άλλο ερώτημα. Έχουμε αυτή τη στιγμή δύο κατηγορίες, δύο περιοχές ε, περιφερειών που πέφτουν στην κατηγορία μεταξύ του 75% και του 90%. Αυτές οι οποίες φεύγουν από αυτή την κατηγορία και αυτές οι οποίες ποτέ δεν είχαν σταθεί σε επίπεδο κάτω του 75% σε κατακεφαλήν ΑΕΠ. Ο στόχος μας είναι να προβλέψουμε έναν τρόπο ισοδίκαιας μεταχείρισης για αυτές τις περιοχές και μπορούμε να φανταστούμε ότι όταν μια περιοχή έχει 80% <clears throat> του μέσου ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης <clears throat> είτε ήταν σε αυτή την κατηγορία προηγουμένως είτε τώρα μπαίνει σε αυτή την κατηγορία η κατάσταση του βιωτικού επίπεδου είναι μία και η αυτή. Και αυτό λέω στον, είπα στον κύριο Ζέμπερ προηγουμένως ότι αυτή τη στιγμή το κατακεφαλήν ΑΕΠ είναι ο κύριος γνώμονας, αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι υπάρχουν και άλλοι δείκτες οι οποίοι μας δίνουν μια καλύτερη εικόνα της κατάστασης μιας περιφέρειας. Όταν όμως έχουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο κατακεφαλήν ΑΕΠ οι περιφέρειες αυτές, αυτό θα πρέπει να οδηγήσει και σε μια ίση μεταχείριση. Έχουμε 500 εκατομμύρια κατοίκους στην Ευρώπη, 300 εκατομμύρια από αυτούς βρίσκονται στις λεγόμενες περιοχές του phasing out και 30 εκατομμύρια βρίσκονται σε περιοχές οι οποίες δεν εμπίπτουν στη χρηματοδότηση. Δεν μιλάμε για λίγο τμήμα του πληθυσμού επομένως μάλλον 30% σε περιοχές του phasing out και 30% σε περιοχές που δεν χρηματοδοτούνται. Είναι συνολικά ένα 60 εκατομμύρια ατόμων, είναι πάνω από 10% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και αυτό το ποσοστό του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ένα θετικό τρόπο. Και επομένω έχουμε μια θετική αντιμετώπιση <clears throat> για την αντιμετώπιση και αυτών των κατηγοριών. Η στοχοθεσία μας είναι να μειώσουμε τις, ε, τις ανισότητες και αυτό θα πρέπει να γίνεται επί τη βάση του επίπεδου των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι διάφορες περιοχές. Η πρότασή μας θα είναι οι περιοχές μετάβασης να αντιμετωπίζονται μέσα στην <clears throat> περίοδο προγραμματισμού με τον ίδιο τρόπο. Εάν βρίσκονται στη διαδικασία του phasing out, τη εξόδου δηλαδή από μια κατηγορία χρηματοδότηση, θα πρέπει να έχουν περισσότερη χρηματοδότηση στην αρχή και λιγότερη στο τέλο, ώστε να γίνεται η λεγόμενη ομαλή προσγείωση. Ε, ενώ οι περιοχέ οι οποίε είναι στην αντίθετη διαδικασία του phasing in θα πρέπει να παίρνουν λιγότερη χρηματοδότηση στην αρχή, περισσότερη στο τέλο, αλλά μέσα στην χρονική αυτή περίοδο των 7 χρόνων να παίρνουν συνολικά την ίδια χρηματοδότηση όπως και οι άλλες. Το θέμα του Εράσμους για τους τοπικούς άρχοντες. Αυτό προβλέπεται στον τρίτο πυλώνα. Ε, υπάρχει και μία παρεξήγηση ορισμένες φορές. Εμείς προσπαθούμε και με τη συνεργασία της Επιτροπής των Περιφερειών να ξεκινήσουμε να υπάρξει αυτή η περαιτέρω εκπαίδευση, η ανταλλαγή των τοπικών αρχόντων ώστε να υπάρχει ένα είδος ε, προγράμματος ε, Εράσμους, αλλά και εκεί θα πρέπει να αποχωρήσουμε σταδιακά. Για τα θέματα του αθλητισμού, θα σας δώσω μια αθλητική απάντηση. Ναι, θα πρέπει να προβλεφθεί αυτό και αυτό εξαρτάται από τις διάφορες χώρες, αν μέσα στα προγράμματά τους θέλουν να έχουν μια τέτοια αντιμετώπιση. Είχαμε και καλές εμπειρίες από προγράμματα όπως αυτό το οποίο ήταν το ειδικό πρόγραμμα για τη Βόρεια Ιρλανδία και αυτά τα προγράμματα έχουν συμβάλει τα μάλα για να υπάρξει και βελτίωση της ε, γενικής κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης μέσω των ε, επενδύσεων στον αθλητικό τομέα. Κύριε Άλβες, νομίζω ότι μιλάτε για τον κανονισμό νη συν δύο, έτσι δεν είναι. Όχι κύριε Επίτροπε. Πρόκειται για την αιρεσιμότητα και την εφαρμογή της της ε, χρηματοδοτήσεις των διαδοτικών ταμείων προς τις περιφέρειες. Λέει ο κύριος Άλβες. ναι, η αιρεσιμότητα φυσικά θα πρέπει να εφαρμόζεται στο Περιφερειακό Ταμείο αλλά με τη μορφή που έχει συμφωνηθεί με τις περιφέρειες. Ποιες προϋποθέσεις είναι αυτές οι οποίες θα συμφωνηθούν και θα πρέπει να επιτευχθούν στην πράξη για να μπορεί να υπάρχει μια επιταχυμένη εφαρμογή των ταμείων και να αντιμετωπίσουμε τις καθυστέρησεις που βλέπουμε σήμερα. Η εδαφική συνεργασία θα πρέπει να ενισχυθεί για τις μακροπεριφέρειες δεν προβλέπεται να υπάρξει πρόσθετη χρηματοδότηση Απλώ ο στόχος των μακροπεριφερειών είναι να υπάρξει μια καλύτερη μορφή συντονισμού και συνεργασίας η οποία μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη, στη βέλτιστη χρησιμοποίηση των υπαρχόντων πόρων. Οι περιφέρειες οι οποίες είναι αστικού χαρακτήρα, κύριε Βόν, οι αστικοί χώροι. Εμείς έχουμε συζητήσει πολλές φορές το θέμα αυτό δεν έχουμε την πρόθεση να δημιουργήσουμε ένα συγκεκριμένο ταμείο για τις αστικές περιοχές, αλλά μέσα στα υπάρχοντα ταμεία να προβλέψουμε ένα συγκεκριμένο ποσοστό, το οποίο είναι υποσυζήτηση του προϋπολογισμού, το οποίο θα είναι προσδιορισμένο για τις αστικές περιοχές. Βέβαια, εναπόκειται στα κράτη-μέλη να αποφασίσουν τι τι θεωρούν μεγάλες αστικές περιοχές. Για κάποια κράτη 100.000 πληθυσμός μιας πόλης θεωρείται ήδη ότι δημιουργεί μια μεγάλη, ένα μεγάλο αστικό σχηματισμό, ενώ για άλλες χώρες μιλάμε για εκατομμύρια κατοίκων. Επομένως το κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να δημιουργήσει τις δομές που θεωρεί λογικές για την αντιμετώπιση των μεγάλων αστικών περιοχών, αλλά η κατεύθυνση της αντιμετώπισης των αστικών περιοχών θα πρέπει να είναι γενική. Νομίζω και σε πάρα πολλά ταμεία ήδη αντιμετωπίζεται αυτό το θέμα και θέλω να σας ευχαριστήσω για την επικοδομητική συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Επίτροπε για αυτή την μακρά ανταλλαγή απόψεων. Ε, είμαι βεβαία ότι θα πιέσετε το γενικό σας διευθυντή να έρθει στην Επιτροπή μας. Μα του αρέσει, του αρέσει το λέει Επίτροπος έτσι ώστε να ξέρουμε ανα πάσα στιγμή ποια είναι η στόχευσή σας, πώς προωθούνται τα ζητήματα τα οποία συζητούμε εδώ. Σας ευχαριστούμε και πάλι κύριε Επίτροπε.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 Αγαπητοί συνάδελφοι, ήγγει και η ώρα των ψηφοφοριών. Έχουμε πολλές δύσκολες και μακρές ψηφοφορίες, επομένως ετοιμαστείτε, οπλιστείτε με τις κάρτες σας. Να ελέγξουμε πρώτα, να κάνουμε μια δοκιμή ότι λειτουργούν οι κάρτες μας. Να ξεκινήσει λοιπόν ο έλεγχος. Ελέγχουμε λοιπόν, άρχεται η ψηφοφορία, ας πούμε. Ψηφίζουμε, να δούμε αν λειτουργούν οι κάρτες μας. We are closing the vote. Not everybody is yet there, but, but I don't know why. Δεν λειτουργήσαν όλες οι κάρτες από ό,τι φαίνεται. Πάντως πέρασε της ψηφοφορίας. I understand that everybody's machine is working. Ε, λοιπόν, λειτουργήσαν όλες, ε, όλα τα μηχανήματα. Παρακαλώ πολύ ηρεμήστε, ησυχάστε και να ξεκινήσουμε το 13. Ε, έκθεση, ε, συγγνώμη, σχέδιο γνωμοδότησης Λάμπερτ Βαν Νίστερο, Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργούς Γύρανσης. Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε με τον πρώτο συμβιβασμό υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται σαφώς. Συμβιβασμός 2 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Α, ξέχασα τις ε, αποχές, λέει η Πρόεδρος. Συμβιβασμός 3, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. 36 εγκρίνεται. 36 κατά. Αποχές εγκρίνεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε σε θεολογικές σκέψεις τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται. Θα κάνουμε έναν γρήγορο έλεγχο. Τροπολογία 17 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ναι, 23 ψήφοι κατά 18 υπέρ, άρα απορρίπτεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 18 ε, καταπίπτει. Συμβιβασμός 8 υπέρ. 4, ε, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 9 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 10 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 11 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 12, συμβασμός 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Η τροπολογία 27 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 28 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Για την 29 έχουμε ψηφοφορία κατά τμήματα. Έχει, το έχει ζητήσει η κυρία Ντέλη. Πρώτο τμήμα, υπέρ του πρώτου τμήματος λοιπόν της τροπολογίας 29, κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται η ψηφοφορία μας. Πέρας. 39 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά, καμία αποχή εγκρίνεται. Περνάμε τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, σε ένα πολύ δύσκολο θέμα, πολύ δύσκολη ψηφοφορία. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να είστε συγκεκριμένοι, ε, συγκεντρωμένοι συγγνώμη, και πολύ προσεκτικοί. Πρόκειται και για την έκθεση της κυρίας Κουστάντσε Κρέλ. Πολιτικές προκλήσεις και δημοσιονομική πόρη για μια βιώσιμη Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το 2013. Η Κωνσταντσα θέλει να πει δυο λόγια, ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πράγματι, πρόκειται για μια δύσκολη ψηφοφορία. Θα ήθελα λοιπόν πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω όλους όσους ε, ε, με πολύ δραστήριο και ενεργητικό τρόπο ε, εργάστηκαν έτσι ώστε να ολοκληρώσουμε αυτήν την γνωμοδότηση. 103 τροπολογίες υπευλήθησαν και στην ουσία μονάχα μια μισή εβδομάδα είχα στη διάθεσή μου για να συζητήσω με τους συγγραφείς αυτών των τροπολογιών και με τους σκιώδεις ε, εισηγητής ε, γιατί άργησε πολύ η μετάφραση ε, την είχαμε πριν, από πάση περιπτώσει δεν είχαμε τη δυνατότητα να μεταφέρουμε την ψηφοφορία γιατί πρέπει να δώσουμε τη γνωμοδότηση στον κύριο Γκαρίγια τώρα. Κάναμε λοιπόν γρήγορα τις διαπραγματεύσεις, τις συζητήσεις. Εάν είχα δεχτεί και τις 103 τροπολογίες θα είχαμε τότε δημιουργήσει ένα τεράστιο χοντρό βιβλίο το οποίο δεν θα κατανοούσε κανείς. Γι' αυτό λοιπόν ε, στους συμβιβασμούς στους οποίους κατέληξα με τους σκιώδης συγητής ε, προσπάθησα να πω σαφώς ότι στόχος μας είναι να ζητήσουμε από την Επιτροπή ΣΟΥΡΕ ε, να ζητήσουμε σωστό προϋπολογισμό για όλες τις δραστηριότητες και στρατηγικές Συνοχή. Ε, νομίζω ότι αυτό ήταν το κυριότερο σημείο. Δεν υπήρχε λόγος να μπούμε σε τρομέρε λεπτομέρειες. Μετά θα δούμε τι θα κάνουμε με τους αβγ πόρους. Κυρίως έπρεπε να θέσουμε κάποιες αρχές. Και να σας πω ένα παράδειγμα. Στην παράγραφο 5 αναφερόμαστε σε προτεραιότητες. Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να συζητήσουμε. Έχουμε διάθεση συζήτησης. Είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε ε, τροπολογίες για να δείξουμε ότι δεν είμαστε αυτιστικοί, ότι δεν είμαστε περιορισμένοι ε, στα δικά μας θέματα, ότι θέλουμε να προσαρμοστούμε στην πολιτική συνοχής και ότι δεν χρειάζεται εδώ ε, να αναφερθούμε σε τρομερές λεπτομέρειες για, την ε, βιο... για τις βιοκαλλιέργειες, ε, για την βιοπικιλότητα, για τον αθλητισμό, για το ένα, για το άλλο. Ανοιχτή σε κάποιες προθέσεις. Γι' αυτό λοιπόν προσπάθησα να ε, συμπιέσω όλες αυτές τις τροπολογίες σε ένα συμβιβασμό. Προσπάθησα επίσης να αποφύγω τις αντιπαραθέσεις. Βεβαίως υπάρχουν αποκλίνουσες απόψεις στις διάφορες πολιτικές ομάδες και αυτές οι αποκλίσεις διαφαίνονται κυρίως σε δύο θέματα ας πούμε για το εάν θα υπάρξουν μεταβατικοί κανόνες, αν θέλουμε να έχουμε έναν ενδιάμεσο στόχο ή ένα νέο στόχο, τρία, όλα αυτά ε, αναφέρονται και νομίζω ότι διαφαίνονται στις ε, τροπολογίες. Η έναν νεο στοχο τρια ολα αυτα αναφερονται και νομιζω οτι διαφαινονται στις τροπολογιες η σουρε δεν χρειάζεται να ε, ξέρει ποιος κανονισμός θα ισχύσει για ποια περιοχή. Ε, αυτό που θέλουμε εμείς είναι να υπάρξουν, δηλαδή να αναγνωριστεί ότι υπάρχουν περιφέρειες ε, μεταβατικές, σε μεταβατική κατάσταση και ότι θα υπάρξουν κανονισμοί που θα τις διέπουν το πώς, το πότε, το λεπτομεριακό μπορούμε να το δούμε και αργότερα και θα χρειαζόμαστε, θα χρειαστούμε σίγουρα περισσότερο χρόνο και θα πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτές τις λεπτομέρειες αργότερα. Γι' αυτό λοιπόν σας ζητώ να ψηφίσετε τις προτάσεις συμβιβασμού ε, και η περαιτέρω λεπτομεριακή συζήτηση να αφαιθεί λίγο στην άκρη για την ώρα και θα την ξαναπιάσουμε αργότερα. Δεύτερον, είναι απαραίτητο να λύσουμε το θέμα των φόρουμ σκέψης. Ενδεχομένως δεν έγινε απολύτως κατανοητό. Τώρα, κάθε χρόνο μπορεί να μείνουν, να παραμείνουν χρήματα. Πολλά εκατομμύρια βλέπε και δις φυσιολογικά τα χρήματα αυτά επανακατατίθενται στους εθνικούς προϋπολογισμούς και επομένω, ε, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το ίδιο πράγμα τα χρήματα αυτά, θα χρησιμοποιηθούν για κάτι άλλο. Στις προτάσεις τροπολογιών που έχουν υποβληθεί υπάρχουν ε, διάφορες ε, προτάσεις να χρησιμοποιηθούν στο ίδιο κράτος μέλος, να χρησιμοποιηθούν στην ίδια περιφέρεια, να ξαναμπούν στο προπολογισμό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εδώ έχουμε κάνει συμβιβαστική πρόταση. Ακολουθήστε την παρακαλώ γιατί τα χρήματα αυτά, οι πόροι αυτοί θα πρέπει να παραμείνουν στον προϋπολογισμό ε, της συνοχής δεν πρέπει να επανέλθουν, να επανακατατεθούν στους εθνικούς προϋπολογισμούς. γιατί αυτό είναι ένα σημείο τριβής ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο και τις χώρες μέλη οι Υπουργοί Οικονομικών των Κρατών Μελών θέλουν να ξαναπάρουν πίσω τα χέρια, τα χρήματα αυτά. Και νομίζω ότι κάτω από τις συνθήκες που ισχύουν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πολύ καλά τα χρήματα στον προϋπολογισμό και πρέπει να κερδίσουμε αυτή τη μάχη προτού περάσουμε στην μεγαλύτερη ε, διαμάχη για, το μέλλον. Γι' αυτό σας ζητώ να υποστηρίξετε αυτή τη συμβαστική λύση. Μερικές φορές δεν έχω φέρει ακριβώς αυτά που λέει επιλέξει η κάθε τροπολογία στη συμβαστική τροπολογία. Προσπαθώ να μεταφέρω το πνεύμα της κάθε τροπολογίας για να διευκολύνουμε την ε, ψηφοφορία. Και θα κάνω και μια προφορική τροπολογία σε, σε κάποιο σημείο για να υπάρξει καλύτερη ε, διευκρίνηση της παραγράφου 19. Υπήρξε και ένα πρόβλημα με τη μετάφραση και νομίζω ότι δεν είναι κάποια δυσκολία, μπορούμε κάπως να το ξεκαθαρίσουμε. Ε, φυσικά η γνωμοδότησή μου δεν έχει σαν στόχο να τροποποιήσει τις συνθήκες. Όσο ισχύει η συνθήκη, η υποστήριξη των υπερπεριφερικών περιοχών μέσω του Ταμείου Συνοχής θα εξακολουθήσει να υφίσταται. Και έχω καταθέσει μια έχω θεωρήσει το ότι να υπάρξει μια τροπολογία για το θέμα αυτό ως υπερβολική και ως περιττή γιατί υπάρχει ήδη αυτή η ρήτρα στις ε, συνθήκες. Μην θέσετε λοιπόν και άλλες τροπολογίες αυτού του είδους. Κατά τα άλλα σας εύχομαι καλή τύχη. Ευχαριστώ. Ε, δεν ήξερα ότι θα μιλήσεις ε, τόσο πολύ. Λαμπέρ, ελπίζω να μην μακρηγορήσεις και εσύ τόσο πολύ. Κοιτάξτε, λέει ο κ. Βανίστερόι, ε, πρόκειται για μια ε, ιδιάζουσα έκθεση που έρχεται σε μια ιδιάζουσα στιγμή. Δεν έχουν προετοιμάσει όλες ε, οι επιτροπές τόσο ενδελεχείς γνωμοδοτήσεις προς την ΣΟΥΡΕ. Εμείς ε, είχαμε μία πλήρη συζήτηση και πιστεύω ότι έτσι έπρεπε να έχει γίνει και έχουμε τώρα μία πλήρη γνωμοδότηση την οποία θα την υποβάλουμε ε, στην συγκεκριμένη περίπτωση την 10η Φεβρουαρίου. Και νομίζω ότι θα πρέπει να υπεραμεινθούμε των στοιχείων ε, τα οποία συζητήσαμε εδώ. Made by, ε, rapporteur. Ακούσαμε λοιπόν προσεκτικά την εισηγήτρια σχετικά με αυτά τα σημεία τα οποία, επί των οποίων ήθελε να επιστήσει την προσοχή μας και γιατί δεν ήταν αρκετά σαφή έχω την αίσθηση ότι όσον αφορά ας πούμε τους μεταβατικούς ε, κανόνες ή αυτές τις μεταβατικές ε, κατηγορίες υπάρχουν ε, κάποιες νέες πληροφορίες που ακούσαμε σήμερα το πρωί διαστόματος του Επιτρόπου. και μέσω της ε, γραμματείας ε, νομίζω ότι θα πρέπει να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να μην διονυστεί αυτή η συζήτηση και να βρουν τη θέση τους ε, τα στοιχεία αυτά στην συζήτησή μας. Πάντως νομίζω ότι είναι απολύτως απαραίτητο να έχουμε επιπλέον συζήτηση για αυτά. Πέρα όμως από αυτό που λέω τώρα, πρέπει να πω ότι για τη συγκεκριμένη ψηφοφορία το ΕΛΚ συμφωνεί με τους συμβιβασμούς. Σε αυτή τη φάση αυτό πρέπει να κάνουμε. Uh, uh, uh, Έχουμε ένα πρόβλημα σχετικά με τους έχοντες δικαίωμα ψήφου. Και στο ΕΛΚ και στους σοσιαλιστές από ό,τι μου λένε. Οι πράσινοι όχι, είναι καλά παιδιά. Λοιπόν, ίσως χρειαστεί να διορθώσουμε λίγο το αποτέλεσμα. Λοιπόν, θα προχωρήσω στην ψηφοφορία αυτή με πολύ αργό ρυθμό, έτσι ώστε να μην υπάρξουν λάθη να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, συμβιβασμός 1 υπέρ κατά σαφές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 8 Υπάρχει επ' αυτού προφορική τροπολογία. Είναι κανείς κατά της προφορικής τροπολογίας. Όχι. Επομένω ψηφίζουμε την τροπολογία 8 έτσι όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ. Κατά. Αποχέ εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 11. Και στην τροπολογία 11 υπάρχει προφορική τροπολογία που έχει ζητηθεί από την κυρία Ματσόνη. Ε, είναι κανείς ε, κατά. Α, δεν ψηφίζουμε λοιπόν την προφορική τροπολογία. Θα ψηφίσουμε όμως την αρχική ε, τροπολογία 11 υπέρ. Κατά. Αποχέσε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 12 υπέρ. Τροπολογία 12 υπέρ. Α, ναι, ναι. Να σταματήσουμε για λίγο. προφορική τροπολογία επί της τροπολογίας 11. Από ό,τι άκουσα, είπατε ότι δεν έγινε δεκτή η προφορική τροπολογία. Ναι, ναι, ναι. Δεν έγινε δεκτή η προφορική τροπολογία. Ναι, ποιος καταψήφισε. Η Κωνσταντζα. Εντάξει. Εντάξει, όχι, δεν θέλω έλεγχο. Απλώς ήθελα να αποσαφηνίσουμε τα πράγματα. Τροπολογία 12. Υπέρ. Υπέρ, κατά, αποχές νομίζω πως εγκρίνεται αλλά κάποιοι λένε ότι δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα ε, λοιπόν ελέγχουμε ηλεκτρονικός έλεγχος άρχεται η ψηφοφορία από της τροπολογίας 12 πέρασε 23 υπέρ 17 κατά εγκρίνεται τροπολογία 13 υπέρ κατά. Νομίζω ότι και εδώ πρέπει να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Τροπολογία 13 άρχεται η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας τη ψηφοφορίας. 24 ψήφοι υπέρ 16 κατά, επομένως εγκρίνεται. Συμβιβασμός 3. Υπέρ. Κατά. Ε, αποχές εγκρίνεται. Συμ... Δεύτερο τμήμα της ε, τροπολογίας 14. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 14 υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβασμός 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 5 υπέρ. Εγώ είχα ζητήσει να κάνω μια τροπολογία. Στο σημείο 5 της συμβαστικής τροπολογίας αναφέρονται οι περιοχές οι οποίες έχουν μόνιμα μειονεκτήματα φυσικής προέλευσης. Πρέ νομίζω ότι εδώ πέραν αυτών θα πρέπει να αναφερθούν και οι υπερπεριφερειακές ε, περιοχές οι οποίες δεν καταγράφονται σε αυτή την ε, παράγραφο. Είναι κανείς κατά αυτής της προφορικής τροπολογίας? Είστε κατά της προφορικής τροπολογίας, μάλιστα. Άρα δεν μπορούμε να ψηφίσουμε την προφορική τροπολογία αυτή. Δυστυχώς δεν μπορούμε, άρα ψηφίζουμε το συμβιβασμό 5 χωρίς τη δική σας προφορική τροπολογία. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 43. 43 λοιπόν υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τη 43 άρχεται η ψηφοφορία. The vote is ψηφοφορίας. 26 υπέρ 15 κατά, επομένως εγκρίνεται. Τροπολογία 46 υπέρ, υπέρ της 46 κατά, αποχές, απορρίπτεται. 48 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 6 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 62 Κατά τμήματα η ψηφοφορία, συνάδελφοι, ψηφίζουμε το 62 τμήμα πρώτο, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα της 62, υπέρ, κατά. Μάλλον απερίφθη. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Δεύτερο τμήμα της τροπολογίας 62. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 26 κατά 15 υπέρ, αλλά απορρίπτεται το δεύτερο βήμα της 62. Συμβιβασμός 9 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 10 υπέρ, κατά, αποχές 72 τροπολογία 72 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 73 με προφορική ερώτηση. Είναι κάποιος κατά της προφορικής τροπολογίας επί της 73. Όχι, επομένως ψηφίζουμε την 73 όπως έχει τροποποιηθεί υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 74 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 11 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 53. Έχουμε εδώ έτοιμα για χωριστή ψηφοφορία και ψηφίζουμε μονάχα το δεύτερο τμήμα της 53. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε τώρα το τρίτο τμήμα της 53. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Θα ψηφίσουμε λοιπόν ηλεκτρονικά για το τρίτο τμήμα της 53. Άρχεται η ψηφοφορία. The vote is closed. Πέρας ψηφοφορίας 22 υπέρ 17 κατά επομένως εγκρίνεται. Τροπολογία 75 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 12 υπέρ κατά αποχές το αποτέλεσμα δεν είναι σαφές λοιπόν ηλεκτρονικός έλεγχος για το συμβιβασμό 13 άρχεται η ψηφοφορία πέρας 18 υπέρ 21 κατά καμία αποχή, δύο αποχές συγγνώμη επομένως απορρίπτεται δηλαδή απορρίψαμε το συμβασμό 13 λέει η πρόεδρος άρα πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 78 τροπολογία 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Συμβιβασμός 13. 14. 13. Υπέρ, κατά. Uh, uh, Νομίζω ότι υπάρχει μια προφορική τροπολογία γιατί ώστε να διευκολυθούν τα πράγματα. Εγώ θέλω το level off, αυτή η διατύπωση, να απαλληφθεί. Όχι, όχι, συγγνώμη, έκανα λάθος, αναφερόμουν στο συμβασμό 14, συγγνώμη. Ναι, ναι, ξεχάστε αυτό που είπε. Ψηφίζουμε το 13. Συμβασμό 13. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβασμός 14. Και εδώ έχουμε δύο χωριστές ψηφοφορίες ή όχι. Α, εδώ θέλετε να υποβάλλετε κάποια... Ακούστε προσεκτικά, συνάδελφοι. Θα δείτε ότι στο συμβιβασμό υπάρχει το επίπεδο της συγχρηματοδότησης, τα αγγλικά level of co-financing. Έτσι ώστε ε, ας πούμε στο συμβιβασμό, ε, έτσι ώστε στη συγχρηματοδότηση να μπορεί ας πούμε η Βουλγαρία να πληρώνει 15%. Εν πάση περιπτώσει διαγράφουμε την έκφραση level of και ο συγγραφέας της τροπολογίας συμφώνησε μαζί μου. Ελπίζω λοιπόν να συμφωνήσει και το ΕΛΚ με αυτή την προφορική τροπολογία που διευκολύνει λίγο την κατάσταση γιατί πλέον δεν είναι απαραίτητο να έχουμε ε, ψηφοφορία κατά τρία τμήματα, θα έχουμε ψηφοφορία κατά δύο τμήματα. Είναι σαφές λοιπόν ότι μιλάμε μόνο ε, για συγχρηματοδότηση και όχι επίπεδο συγχρηματοδότησης. Μένει μόνο το co-financing και διαγράφεται το level off. Ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν το πρώτο τμήμα και το τρίτο τμήμα του Συμβασμού 14 και όχι το δεύτερο. Σουέτερ. Θα ψηφίσουμε επί, επί του Συμβασμού 14 χωρίς χωριστή ψηφοφορία, αλλά δεν θα ψηφίσουμε για αυτό το level off. Um Συγγνώμη. Οι πράσινοι δεν είναι οι μόνοι οι ζήτησαν ψηφοφορία σε τμήματα. Αν μπορούσε και η ομάδα των συντηρητικών να αποσύρει την δική τους ε, αίτηση για χωριστή ψηφοφορία, θα ήταν καλό γιατί έτσι θα γλιτώσουμε την τρίτη ψηφοφορία στο τρίτο τμήμα. Ναι, αλλά ίσω είναι ασφαλέστερο να ψηφίσουμε ε, όπως ήταν αρχικά με χωριστή ψηφοφορία. Ε, να ψηφίσουμε λοιπόν το πρώτο και το τρίτο τμήμα. Υπέρ του πρώτου τμήμα του συμβιβασμού 14. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τρίτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 87. Τροπολογία 87 υπέρ. Κατά. Επαλήθευση για την τροπολογία 87. Το αποτέλεσμα δεν είναι σαφές. Άρχεται η ψηφοφορία. Έληξε η ψηφοφορία. 22 υπέρ, 22 κατά, ισοψηφία. Άρα απορρίπτεται. Συγγνώμη, απορρίπτεται. Συμβαστική τροπολογία υπαριθμό 15. Ψήφι Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 90. Ψήφι Κατά. Αποχές δεκτή. 91. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 95 έχουμε προφορική τροπολογία ποιος είναι κατά της προφορικής τροπολογίας ψηφίζουμε τα 95 όπως τροποποιήθηκε υπέρ κατά αποχές δεκτή περνάμε στη συμβαστική τροπολογία υπέρ 16 ψηφί κατά αποχές δεκτή. Στην παράφο 19 έχουμε μια προφορική τροπολογία. Θέλ, το Στάντσα θέλει κάτι να πει. Ναι, αυτή η παράγραφος ε, υπαριθμών 19 είναι ένα ζήτημα το οποίο συζητείται ακόμα και σε επίπεδο μεταφραστικό, δηλαδή μετάφρασης ε, του κειμένου τη Πασμού 19. Η τροπολογία 102 έχει συμπεριληφθεί και τονίζεται ιδιαίτερα το γεγονό ότι η πολιτική συνοχή που ε, είναι ευφυής, περιβαλλοντική, ανοιχτή σε όλους κλπ. Είναι ένας τρόπος για βοηθάει στην εφαρμογή της στρατηγικής 2020 και τονίζεται ότι αυτή είναι μια απόδειξη σχετικά με την σημασία της ε, πολιτικής συνοχής και απορρίπτει κάθε κατακαιρματισμό αυτής της ε, πολιτικής στις, ε, στον προπολογισμό και στις γραμμές αυτού. Και... Αυτό έχει συζητηθεί και συμφωνηθεί με όλους τους συντάκτες τροπολογιών και τους χειόδης συζητητές και νομίζω ότι είναι μια λογική συμβαστική λύση. να αποφεύγουμε έτσι την παγίδα στην οποία μπορούμε να πέσουμε. Λοιπόν, τι ψηφίζουμε τώρα. Ψηφίζουμε την παράγραφο 19 όπως τροποποιήθηκε από την Κωνσταντζα μόλις το λέω τώρα. Ψήφι πέρα. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Και τώρα θα περάσουμε στην τελική ψηφοφορία. Ηλεκτρονικός παρακαλώ. Άρχεται ψηφοφορία. πέρα της ψηφοφορίας. 41 ψήφοι υπέρ, μία ψήφος κατά και μία αποχή. Καλό το αποτέλεσμα, δεν λέω. So now we move, uh, dear colleagues... Αγαπητοί συνάδελφοι, θα εορτάσουμε αργότερα, αλλά τώρα είμαστε στο επόμενο σημείο της Μεσαίας Διατάξεως. Είναι η έκθεση του συνέλφου Κόβατσετς ε, για την στρατηγική ε, σχετικά με τους Ρώμα. Περνάμε με, ε, στην ψήφιση της συμβαστικής τροπολογίας υπαριθμών 1, ψήφι υπέρ, κατά, εποχές, δεκτή. Και τώρα περνάμε στην τροπολογία υπαριθμών 2, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Τροπολογία 11, η οποία τροποποιήθηκε προφορικός. Υπάρχει κάποιο που θα είναι κατά τη προφορική τροπολογία. όχι. Ψηφίζουμε την 11 όπω έχει τροποποιηθεί, ψηφι υπέρ. Κατά. αποχέ. Θα πρέπει να επαληθεύσουμε. Τροπολογία 11, ψήφι υπέρ. Ε, συγγνώμη, ψηφορία πέρα της ψηφοφορίας και απορρίφθηκε 25 ψήφοι κατά 18 ψήφοι υπέρ και μία αποχή. Περνάμε στην τροπολογία 12 ψήφοι υπέρ κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 13 Α, συγγνώμη, καταπίπτει. Περνάμε στην φασιστική τροπολογία 3. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία υπερθμών 24 ψήφι υπέρ. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική πρόταση 24 ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τροπολογία 27 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, δεκτή. 28 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 29 έχουμε προφορική τροπολογία είναι κανείς κατά της προφορικής τροπολογίας όχι ψηφίζουμε την 29 όπως τροποποιήθηκε ψηφί κατά αποχές δεκτή περνάμε στην 31 ψηφί κατά τώρα κατά ας επαληθεύσουμε καλού κακού 31. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία, 22 ψήφοι υπέρ, 18 κατά, δεκτή. Ε, συμβαστική πρόταση 5 ψήφοι υπέρ. Κατά. Αποχές ε, δεκτή. Συμβαστική τροπολογία 6. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 40. Α, είναι ταυτόσιμη. Δεν ψηφίζουμε. Περνάμε στην συμβασμό 7. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Περνάμε στην τροπολογία 44. Καταπίπτει. μου είπαν ότι καταπίπτει. Περνάμε στην 49. Ψήφι υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 50. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Στην 51 υπάρχει μια προφορική τροπολογία. Αντιτίθεται κανείς στην προφορική τροπολογία ψήφι υπέρ της 51 όπως βίντεο Κατά αποχές εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε επί του συνόλου της νομοδοτήσεως όπως τροποποιήθηκε ψήφι υπέρ. Πέρα ψηφοφορίας. 39 ψήφι υπέρ, μία ψήφος κατά, τέσσερις αποχές, συγχαρητήρια. Αγαπητοί συνάδελφοι, συγγνώμη, ο Βίκτο θέλει να πει κάτι το σημαίνον. Κυρία Πρόεδρε. Εκφράζω τη λύπη μου για το γεγονός ότι ορισμένε φορές η πολιτική μας τοποθέτηση συγκρούεται με τις ευρωπαϊκές μας αρχές. Γιατί η προφορική μου τροπολογία έλεγε ακριβώς αυτό το οποίο είχε πει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάτι επανάληψη. Αυτό το οποίο έχει αναφέρει και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εγώ θυμάμαι αυτά που είπε η κυρία Ρέντινγκ. Φτάνει. Αρκετά είναι αρκετά. Και βλέπω τώρα η διάκριση να γίνεται ευρωπαϊκή αξία. Θέλω να καταγραφεί αυτό στα πρακτικά παρακαλώ. Πάμε στο σημείο 6 της μέσης διάταξης που είναι η γνωμοδότηση του Σαλβατόρε Καρόνα για την Ευρώπη ως πρώτο τουριστικό προορισμό στον κόσμο. Αγαπητοί συνάδελφοι, μην φύγετε ή μάλλον αυτοί οι οποίοι θέλουν να φύγουν να πάνε σε τουριστικούς προορισμούς, ας φύγουν χωρίς φασαρία. Δεν κάνουμε διάλειμμα. Όλμπερτ και Ολεϊνίτσα, άμα θέλετε να μιλήσετε εκτός της αιθούσης, παρακαλώ. Ο Σαλβατόρε Καρόνα έχει το λόγο. Πολύ σύντομα, Πρόεδρε, διότι η έκθεση αυτή εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Μεταφορών και γιατί η πρόταση της Επιτροπής πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση για να δώσει μια νέα όθηση σε έναν κλάδο αυτόν του τουρισμού που είναι όχι μόνο ζωτική συμφίση για τις οικονομίες μας αλλά και συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της εικόνας ε, της Ευρώπης ανά τον κόσμο. Ως εκ τούτου θεωρώ πως η πρόταση της Επιτροπής αποτελεί μια καλή βάση, πιστική βάση, επί της οποίας μπορούμε να οικοδομήσουμε μια ανανεωμένη πολιτική του τουρισμού τα προσεχή έτη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση σήμερα είναι ο πρώτος τουριστικός προορισμός ε, στον κόσμο. Το 2008 κατεγράφησαν πάνω από 370 εκατομμύρια αφήξεις περίπου το 40% του συνόλου των αφήξεων ανά τον κόσμο και στο πρώτο εξάμεινο του 2010 τα στοιχεία δείχνουν μια ανάκαμψη αν και πιο αργή σε σχέση με άλλες περιοχές του κόσμου όπως η Ασία σε σχέση με την κάμψη που είχε καταγραφεί το 2009. Ιδιαίτερα υπάρχει αύξηση των αφήξεων από ορισμένε χώρες όπως η Κίνα, η Ρωσία και η Βραζιλία. Τώρα ο τουρισμός λοιπόν είναι μια οικονομική δραστηριότητα σε θέση να, προκαλέσει ανάπτυξη και απασχόληση και περίπου 2 εκατομμύρια επιχειρήσεων που καλύπτουν το 5,2% της συνολικής απασχόλησης στην Ευρώπη. Ο κλάδος του τουρισμού δημιουργεί πάνω από 5% του ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόκειται για ένα ποσοστό το οποίο συνεχώς δεν είναι ευξανόμενο. Το τομέας του τουρισμού συμβάλλει αποφασιστικά στην ε, ανάπτυξη και της ε, οικονομίας και της κοινωνίας, ιδιαίτερα στις ε, περιοχές της υπαίθρου, στις ορνές περιοχές, στις παράκτης περιοχές, στις νησιωτικές και στις περιφερειές εξού η ανάγκη να υπάρξει μια ευρωπαϊκή πολιτική τουρισμού ε, για να υπογραμμίσουμε τις ε, ιδιαιτερότητες ε, κάθε κράτους μέλους μέσω όλο και μιας μεγαλύτερης ολοκλήρωσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό το πλαίσιο Αποφασιστική σημασία έχει ο ρόλος των περιφερειών και των δήμων κοινοτήτων που θα πρέπει να είναι σε θέση να δυναμωτήσουν έναν ρόλο όλο και πιο ενεργό και να πρωταγωνιστήσουν με μια εμπλοκή στην κατάρτιση μιας νέας πολιτικής τουρισμού. Οι ανάγκε που κατέθεσε ε, προτεραιότητα ε, η Επιτροπή για μια στρατηγική πολιτική υπέρ της ανάπτυξης ε, του τουρισμού στην Ευρώπη μπορούν να συνοψιστούν σε δύο ώρες, σε δύο ώρες ανταγωνιστικότητα και βιωσιμότητα, εφορία. Και σε ευθεία γραμμή με τη συνθήκη της Λισαβόνας η Ευρωπαϊκή Πολιτική Τουρισμού στοχεύει ιδιαίτερα στο να παροτρύνει την ανταγωνιστικότητα του κλάδου χωρί όμω να ξεχνάμε ότι θα πρέπει να υπάρξει οικονομική ανάπτυξη και αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί δίχως ε, την αηφορία του κλάδου. Η γνωμοδότησή μου επικεντρώνεται σε αυτά τα δύο κεντρικά θέματα. Δηλαδή η Ευρώπη να μπορέσει να διατηρήσει την θέση της ε, ως ε, παγκόσμιος ε, προορισμός του τουρισμού και να εμπλουτίσει την, και να τονίσει την διαφορετικότητα και την ποικιλομορφία των περιφερειών της. Η Ευρώπη χρειάζεται να προτείνει μια προσφορά ε, τουρισμού ε, κάνοντας, ε, δίνοντας βάση στον πολιτισμό της, στην ιστορία της κλπ. Παράλληλα προστατεύοντας το περιβάλλον, τη συνεχή κατάρτιση των αποσχολημένων στον κλάδο, η ενίσχυση των μεταφορών, η ανταλλαγή των πρακτικών μεταξύ των 27 κρατών μελών της Ένωσης, έναν καλύτερο συντονισμό των εμπλεκομένων στον τουριστικό τομέα κάνοντας λοιπόν αυτό το νέο ποιοτικό άλμα στον ε, κλάδο. Στο σχέδιό μου αναφέρεται το δυναμικό της Ευρώπης στον τομέα ε, αυτό, οι επιπτώσεις στην οικονομική, κοινωνική και εδαφική ε, συνοχή και θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσπάθειά ε, μα σε μέτρα τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την Να Αναφέρουμε στην βελτίωση τη προσφορά, τη διαφοροποίηση των παραχών υπηρεσιών και αγαθών και την στήριξη νέων μορφών τουρισμού που ξεπερνάνε το πλαίσιο της ε, εποχικότητας και να προωθήσουμε περαιτέρω την κατάρτιση των ε, απασχολουμένων στον κλάδο. Υπάρχουν και κάποιες άλλες πτυχές που έχουν πολύ μεγάλη σημασία, αλλά για λόγους ε, ε, ε οικονομίας δεν μπόρεσα να αναπτύξω, όπως η πρόθεση προγραμμάτων για επιχειρήσεων που δραστηριοποιούν το κλάδο, μια εφαρμογή της οδηγίας για το ηλεκτρονικό εμπόριο που θα πρέπει να εφαρμοστεί στον τομέα αυτό. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Φυσικά προσβλέπω στις ε, παρατηρήσεις σας, στα σχόλιά σας που δίχως άλλο θα βελτιώσουν αυτό το σχέδιο νομοδότησης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ λέει η Πρόεδρος. Έχουμε τους σκιώδεις εισηγητές. Θέλετε να λάβετε τον λόγο. Ναι, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Συμμεριζόμαστε σε γενικές γραμμές την άποψη του εισηγητή στο γεγονός ότι πρέπει να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού τουρισμού και θα πρέπει να ενισχυθεί και η αηφορία του κλάδου αυτού. Είναι προφανές λοιπόν ότι όλες οι προσπάθειες που καταβάλλονται στα επίπεδα της καινοτομία είναι πολύ σημαντικές για να ανυψωθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Υπήρου. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον καθαρά εποχιακό το χαρακτήρα, και να ενισχύσουμε τη διαφοροποίηση του τομέα αυτού και φυσικά να στοιχηματίσουμε πάνω στην ποιότητα. Έχουμε καταθέσει μια σειρά από τροπολογίε, μάλλον θα καταθέσουν μια σειρά τροπολογίε σε σχέση με την έκθεση αυτή, για να συμβάλλουμε στη βελτίωσή τη. Πρώτα απ' όλα, έχουμε την εξή σκέψη να αναφέρουμε. Σεβόμενη τη αρχή τη επικουρικότητα, θα πρέπει να αποφύγουμε υπερβολική ρύθμιση στο ευρωπαϊκό έδαφο για τον τουρισμό. Έχουμε βέβαια τις αρμοδιότητες τις οποίες μας δίνει η Συνδίκη της Λισαβόνας, αλλά θα πρέπει να περιοριστούμε σε αυτές. Χρειαζόμαστε επίσης μια πολιτική ανταγωνισμού που θα εξασφαλίσει την υγεία του τομέα και θα ξεπεράσει την κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης παραδείγματο χάρη στην Ισπανία, στι Βαλεαρίδε από την Τόμα Κουκ που γνωρίζει πολύ καλά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Πρέπει να υπογραμμίσουμε λοιπόν την ανάγκη της πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των άλλων επιχειρηματιών σε χρηματοδότηση, ιδίω μικροπιστώσεις και την ανάγκη να συνεχίσουμε να επεξεργάζομαστε ε, προγράμματα επανορθωτικού χαρακτήρα όπως είναι το Καλύψο και να σκεφτούμε για προγράμματα ανταλλαγής τουριστών μεταξύ κρατών μελών στην χαμηλή σεζόν το οποίο θα βοηθήσει την τουριστική δραστηριότητα ιδίως για τα άτομα τρίτης ηλικίας και επίσης θέλουμε να αποφύγουμε τις επικαλύψεις ε, σημάτων ποιότητος, γιατί υπάρχουν ήδη αρκετά σήματα αυτού του είδους και αν θέλουμε να έχουμε μια ετικέτα ποιότητος στον τουρισμό, να εξετάσουμε με δημοσκοπήσεις την αξία και το αντίκτυπο που θα έχουν τέτοιες ετικέτες. Επίσης έχουμε μία ε, τροπολογία σε σχέση με την αίτηση της Κομισιόν να υπάρχει ένας τουρισμός παράκτιος ο οποίος είναι αηφόρος και βιώσιμος είναι μέσα στα σχέδια της Κομισιόν επομένως μπορούμε να εισαγάγουμε μια τέτοια ε, τροπολογία επίσης πρέπει να δώσουμε και έμφαση στο θέμα των νησιωτικών περιοχών που έχει μεγάλη σημασία ο τουρισμός για αυτές και σε ό,τι αφορά την πρώτη Ευρωπαϊκής Υπήρου ως τουριστικού προορισμού, είναι σημαντικό να υπογραμμίσουμε την επικουρικότητα, να μην υποστηρίξουμε μία περιοχή και όχι μία άλλη, αλλά να υποστηρίξουμε την Ευρώπη σαν σύνολο. Και αυτό είναι σημαντικό γιατί πολλοί έχουν ανησυχίες για την πρόθεση του τουρισμού. Και σε ό,τι αφορά τις αναδυόμενες χώρες, όπως τις λέει η Κομισιόν, Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία και Κίνα, να μπορούμε να έχουμε μια στρατηγική για να προσελκύσουμε τους τουρίστες από αυτές τις χώρες και να τους φέρουμε στην Ευρώπη. Να προωθήσουμε μορφές τουρισμού όπως είναι παραγωγικά ο ιστιοπλοϊκός τουρισμός, ε, ο τουρισμός υπασίας, ο τουρισμός περιοχών που είναι τα κτλ. Και ένα ακόμα θέμα το οποίο είναι σημαντικό. Σε πολλές ε, τουριστικές περιοχές μεγάλης ε, ακτινοβολίας, όπως ήταν οι Βαλεαρίδες χάρη, στην ε, δεκαετία του 1960 υπήρξε άκρατη κατασκευαστική δραστηριότητα. Τώρα πρέπει να ανακτήσουμε αυτές τις υποβαθμισμένες περιοχές και να τις μετατρέψουμε για μία μορφή τουρισμού περισσότερο ποιότητος. Θα πρέπει λοιπόν στις μεροντικές χρηματοδοτικές προοπτικές να υπάρξει και η δυνατότητα ε, αναπροσαρμογής αυτών των περιοχών που είναι πεπαλαιωμένοι η, υποδομή τους για να προσαρμοστούν σε ένα τουρισμό ποιότητας. Λοιπόν, η αναδιάρθρωση επομένως των τουριστικών υποδομών σε αυτές τις περιοχές που είναι υποβαθμισμένες είναι πολύ σημαντικό αυτό και επειδή ο τουρισμός του μέλλοντος βασίζεται στην καινοτομία, στην ποιότητα, στην κατάρτιση κτλ. θα είναι χρήσιμο να συμπεριλάβουμε αυτήν την μνήμα και επίσης να έχουμε μια τροπολογία η οποία υποστηρίζει την, υποστηρίζει την ανάπτυξη των ευρωπαϊκών δικτύων μεταφοράς. Αν δεν υπάρχουν συνδέσεις σε αεροπλάνα, τρένα, πλοία κτλ. Δεν μπορούμε να έχουμε αναπτυγμένο τουρισμό. Πρέπει να τονίσουμε λοιπόν το θέμα αυτό. Έχουμε κάποιον από την, ε, από την ομάδα των φιλελευθέρων, η Ρίκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε εισηγητά, αγαπητοί συνάδελφοι, θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την πολύ καλή του γνωμοδότηση που καλύπτει όλα αυτά τα οποία πρέπει να αναφερθούν. Η κυρία Σάβησάρ είναι η εισηγήτριά μας για το θέμα αυτό, αλλά δεν μπορούσε να έρθει στη σημερινή συνεδρία. Μου ζήτησε να μεταφέρω τις ιδέες. Η κυρία Σάβησάρ θέλει να υπογραμμίσει το ότι είναι απαραίτητο να αντιμετωπίσουμε τον εποχιακό χαρακτήρα του τουρισμού να υποστηρίξουμε μια ευρύτερη δραστηριότητα και ιδίως να ενισχύσουμε τον τουρισμό για τους νέους, για τους ηλικιωμένους και για τα άτομα με προβλήματα κινητικότητας. Κάτι άλλο το οποίο σημαντικό είναι ότι πρέπει να αναπτύξουμε βιώσιμες μορφές τουρισμού και αυτές οι μορφές θα πάρουν προεξάρχουσα μορφή στα επόμενα χρόνια και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το φυσικό και πολιτιστικό κληροδότημα κάθε περιοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να επιτύχουμε λοιπόν αυτού του στόχου πρέπει να τονίσουμε την ποιότητα των υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού. Με περισσότερο τεχνολογικό περιεχόμενο και εθνικά εργαλεία τα οποία μπορούν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες που μας δίνουν οι χρηματοδοτήσεις για την κατάρτιση. Η κυρία Σαββισάρ θεωρεί ότι είναι καιρός να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια ευρωπαϊκή ετικέτα ποιότητας που θα δείχνει την ποιότητα των υποδομών και των υπηρεσιών. Με τον τρόπο αυτό θα ενισχυθεί η εικόνα μας και ο τουριστικός μας τομέας. Ευχαριστώ. Thank you uh, very much. Iligoyen, please. Sí, buenos días. Muchas gracias, señora. Καλημέρα σας, ευχαριστώ πολύ Προέδρε. Να συγχαρώ πρώτα απ' όλα τον συναδελφό μου κύριο Καρόνα για την εξαίρετη σχέδιο γνωμοδότησης και να πω ότι η πρόταση της Κομισιόν πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Θα ήθελα να συμπεριλαμβανθούν νέα, κάποια νέα στοιχεία. Όπως όλοι γνωρίζουμε, το δυναμικό του κλάδου του τουρισμού αντιπροσωπεύει πάνω από 10% του ΑΕΠ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για να αντιμετωπίσουμε την ε, οικονομική κρίση και να βελτιώσουμε την απασχόληση. Για να γίνουν όλα αυτά χρειάζεται να λάβουμε υπόψη ότι ο το... τουρισμός είναι ένας εγκάριστος τομέας και θα χρειάζεται να καλύψουμε τις ελλείψεις που υπάρχουν σε επαγγελματικό επίπεδο για το, οποίο αντιμετωπίζει ο κλάδο, αλλά και τι διάφορε υποδομέ. Θα πρέπει να προωθήσουμε την καινοτομία και την περιφερειακή συνεργασία, αλλά και τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων κλάδων. Κατά την άποψή μου, είναι απαραίτητο να τονίσουμε την σημασία που ο τουρισμός έχει για τις νησιωτικές περιοχές για τις οποίες είναι η βασική μορφή εσόδων. Ο τουρισμός αποτελεί ένα στοιχείο για την οικονομική ανάπτυξη αυτών των πληθυσμό και την... Ε, χρειάζεται να καταπολεμήσουμε τις ε, επιπτώσεις του εποχιακού τουρισμού με κάποιες συγκεκριμένες προσφορές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει τη δυνατότητα να το πετύχει κάτι τέτοιο. Αυτό εξάλλου ζητεί και ο κλάδος ο τουριστικός. Χρειάζεται να υπάρξουν λοιπόν νέα προγράμματα τουριστικά από τον πράσινο τουρισμό τον πολιτισμικό τουρισμό, τον, ε, τον τουρισμό των ε, τρίτης ηλικία κλπ. Συμφέρω με τον εισηγητή ότι θα πρέπει να οργανωθούν δίκτυα και ενώσεις για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι του τουριστικού κλάδου. Τέλος θεωρώ την θετικότατη πρόταση να δημιουργηθεί ένα ευρωπαϊκό σήμα που θα, με τρόπο αυτό θα αναγνωρίζονται τα προϊόντα ποιότητα. Θα είναι λοιπόν καλό να υπάρξει ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών στις χώρες όπως Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα που είναι πρωτοπόροι σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Επόμενος αγορητής. Ο κύριος Κέλλη. Σας ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω τον εισηγητή και τους κοιόδης. Νομίζω μας έχουν δώσει μια πολύ καλή βάση εργασίας για την ανάπτυξη μιας ε, τουριστικής πολιτικής για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε τελική ανάλυση να δημιουργήσουν τη σωστή υποστήριξη για τα θέματα αυτά. Εγώ έρχομαι από το Killarney, από τη Νότια Ιρλανδία, και έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα προβλήματα της εποχιακότητας που αντιμετωπίζουν και άλλες τουριστικές ε, περιοχές και την πρόκληση για να αναπτύξουμε μια σωστή μορφή τουρισμού. Η εποχικότητα μπορεί να αντιμετωπιστεί με διάφορους τρόπους, ιδίως όταν ε, είναι πιο ηλικιωμένος ο πληθυσμός και έχουν ε, οι πολίτες αυτοί περισσότερο ελεύθερο χρόνο με τη συνταξιοδότησή τους, μπορούν να επεκτείνουν την τουριστική σεζόν. Και έχουμε επίση το θέμα τη προσέλκυση χωρών όπω είναι η Ινδία, η Κίνα, η Νότια Αφρική, θα δημιουργήσουν μια παγκόσμια αγορά. Επειδή αυξάνεται το βιωτικό του επίπεδο, είναι φανερό ότι θα θέλουν να ταξιδεύουν περισσότερο. Επομένω, το θέμα του τουρισμού συνδέεται και με την ευκολία παροχή τροξενικών θεωρήσεων για να είναι πιο εύκολο το ταξίδι. Αυτό είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί από εμά. Νομίζω ότι έχουμε την καλύτερη ευκαιρία σε οποιαδήποτε, εναντί οποιασδήποτε άλλη εποχής, με το ίντερνετ να, διαλαμ, να μεταλαμβαδεύσουμε τις πληροφορίες, να πλησιάσουμε πολλούς ανθρώπους και να δημιουργήσουμε τη θέληση να ταξιδέψει κανείς, ιδίως να έρθει στην Ευρώπη που είναι ο κυριότερος τουριστικός προορισμός σε όλο τον κόσμο. Γιατί στην Ευρώπη έχουμε τα πάντα. Η κάθε χώρα έχει κάτι διαφορετικό να δώσει, αλλά εμεί πρέπει να προωθήσουμε την Ευρώπη σαν σύνορο και να πείσουμε τα κράτη-μέλη να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο. Το λέω αυτό για τη χώρα μου. Πέρσι είχε ένα εκατομμύριο τουρίστες λιγότερο και για ένα πληθυσμό 4 εκατομμυρίων καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Υπήρξαν πολλοί λόγοι όπως η οικονομική ύφεση, η ηφαιστιακή τέφρα κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα, και το έχω πει πολλές φορές συνδέεται με το κακό marketing. Πρέπει λοιπόν να βρούμε τρόπους να προωθήσουμε καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ήπειρο και να χρησιμοποιήσουμε τις βέλτιστες πρακτικές για να δούμε πώς χώρες οι οποίες είναι ικανές στο μάρκετινγκ τα καταφέρνουν. Και ξέρω θα έχουμε προς, θα ε, σε λίγο εν καιρό εκλογές, θα αλλάξει η κυβέρνηση, θα αλλάξει ίσως η όλη προσέγγιση για τα θέματα του τουρισμού Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό και να βελτιστοποιήσουμε και μεγιστοποιήσουμε το δυναμικό μας, αλλά επίση και να αγκαλιάσουμε περισσότερο την Ευρώπη. Πρέπει να είμαστε πιο Ευρωπαίοι και θα ωφεληθούμε περισσότερο από το να έχουμε ένα πιο ευρωπαϊκό πνεύμα να παρακολουθούμε τι κάνουν οι άλλες χώρες της Ευρώπης και τι προωθείται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κάτι που θα βοηθήσει όλους και στην Ευρώπη και στη χώρα του καθενός. Τελευταία παρατήρηση, κάτι άλλο, το οποίο είναι τμήμα της στρατηγικής μας 2020, είναι να και θα αναπτύξει τις δυνατότητε του τουρισμού, είναι η έννοια της κινούμενης νεολαίας. Της νεολαίας που πηγαίνει από χώρα σε χώρα που πηγαίνουν σε μια χώρα και μετά θέλουν να επανέλθουν. Γιατί ξέρω ότι αυτοί οι οποίοι έχουν έρθει στις Βρυξέλλες για να σπουδάσουν θέλουν στη συνέχεια να επανέλθουν. Μπορούν να οργανώσουν ομάδες οι οποίες θα πάνε σε μια χώρα σε μια άλλη. Αυτό το πλαίσιο λοιπόν έχει τεράστια δυναμικότητα. Πρέπει να τη χρησιμοποιήσουμε και να κάνουμε την Ευρώπη όχι μόνο τον πρώτο τουριστικό περιορισμό, προορισμό, αλλά ένα προορισμό ο οποίος και στο μέλλον θα είναι σημαντικό και πηγή οικονομικών ωφέλων. Θέλω να ευχαριστήσω πολύ τον εισηγητή και του κοιότητε, λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πραγματικά. Ευχαριστώ Προέδρε. Ε, με αφορμή αυτή την ε, έκθεση θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε ορισμένα πολύ σοβαρά προβλήματα που νομίζω αντιμετωπίζουν συνολικά οι χώρες μας στον τομέα του τουρισμού και το οποίο δυστυχώς δεν, ε, στο οποίο δεν γίνεται απολύτως καμία αναφορά στην, ε, στο σχέδιο ψηφίσματος ε, και εκδηλώνονται κατά τη γνώμη μου πολύ πιο έντονα στις περιφέρειες. Πρώτο ζήτημα. Υποδομή. Ε, συνήθως οι τουριστικές περιοχές είναι υποχρεωμένες να φιλοξενήσουν έναν πολύ μεγαλύτερο αριθμό από επισκέπτες από, τον, από τους κανονικούς κατοίκους. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα ε, είναι, προς, ε, ευπρόσδεκτοι βέβαια οι επισκέπτες, όμως οι υποδομές είναι πάρα πολύ πίσω. Τουλάχιστον στην Ελλάδα σε πολλά νησιά αντιμετωπίζεται ένα τέτοιο θέμα. Ε, και εννοούμε για βασικές υποδομές, όχι μόνο γενικότερες. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Δεύτερο ζήτημα. Δεν ξέρω σε άλλες χώρες τι γίνεται. Στην Ελλάδα όμως είναι πολλές οι ακτές στι οποίε δεν υπάρχει ελεύθερη πρόσβαση. Είναι ιδιωτικές ακτές ή ιδιωτικοποιούνται οι ακτές με αποτέλεσμα να μην μπορούν οι άνθρωποι να πάνε ελεύθερα να κάνουν τον μπάνιο τους, να κάνουν τη τηλεοθεραπεία κτλ. Τρίτο ζήτημα. Άρα ελεύθερες ακτές. Τρίτο ζήτημα. Τουριστικά γραφεία τα οποία κοροϊδεύουν τους πελάτες τους. Έρχονται οι άνθρωποι για διακοπές στην Ελλάδα και μέχρι να τελειώσουν οι διακοπές το γραφείο έχει φαλυρίσει. Δεν ξέρουν πώς να γυρίσουν πίσω. Κολυμπώντας, περπατώντας, πετώντας, τίποτα. Πέμπτο ζήτημα. Υπερκορεσμένες τουριστικές περιοχές. Βεβαίως, να αναπτυχθεί ο τουρισμός δεν είναι κανένας αντίθετος, αλλά όταν και ο τουρισμός εξυπηρετεί το κέρδος, όπως συμβαίνει στη χώρα μου και αλλού, έχετε το παράδειγμα της Κέρκυρας και έχετε το παράδειγμα της Ρόδου, κύριε Πρόεδρε το γνωρίζετε και ελπίζω να μην το γνωρίζουν και πολλοί από εσά, όσοι το γνωρίζουν όμως ξέρετε ότι υπάρχει, υπάρχει ένας υπερπληθυσμός και μια κατάσταση πάρα πολύ δύσκολη. Ε, τέλος, θα ήθελα να ε, επιστήσω την προσοχή σας πολύ συχνά σε άθλιες συνθήκες εργασίας, είτε είναι μεγάλα ξενοδοχεία, είτε είναι κρουαζιερόπλια. Έχουμε περιπτώσεις από νέους ειδικευμένου ή εργαζόμενου οι οποίοι ειδικεύονται στον τομέα του τουρισμού από τη Βουλγαρία, από τη Ρουμανία, από την Τσεχία, από την Πολωνία, οι οποίοι απασχολούνται σε ελληνικές τουριστικές μονάδες με μισθούς πείνας πραγματικά. Νέοι ναι, άνθρωποι με, 10 ευρώ την ημέρα, με 5 ευρώ την ημέρα, τη στιγμή που η μισθή είναι πολύ πιο μεγάλη, στο όνομα της εκπαίδευσης. Ε, και τέλος, κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα, όπως γνωρίζετε, με το θέμα της άρσης του καμποτάζ. Αυτό έχει επιπτώσεις στον τουρισμό κρουαζιέρας. Δεν γίνεται λόγος για αυτό το θέμα ε, στο στο σχέδιο ψηφίσματος. Είναι σημαντικός αυτός ο, ο, τομέας, αλλά με συνθήκες, με πληρώματα κακοπληρωμένα και σε δύσκολες συνθήκες εργασίας τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τελειώνοντας, θα ήθελα να εκφράσω τη λύπη μου για το γεγονός ότι στο σημείο 8, μάλλον είναι λάθος ε, μετάφρασης φαντάζομαι, γίνεται λόγος ότι οι ηλικιωμένοι μπορούν να αποτελέσουν άτομα που αποτελούν αγορά με μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. Πρώτη φορά διαβάζω κείμενο όπου να γίνεται λόγος ότι άτομα αποτελούν αγορά και μάλιστα με προοπτικές ανάπτυξης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Thank you. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ θα πάρω το λόγο στο όνομα του ε, εισηγητού μας, του σχέδιου εισηγητού, του κ. Τριμόπουλου, ο οποίο δυστυχώ αναγκάστηκε να φύγει. Ε, για μα ο τουρισμό βεβαίω είναι πάρα πολύ σημαντική δραστηριότητα, η οποία ε, αντιπροσωπεύει πολύ μεγάλο ποσοστό θέσεων εργασία και κατέχει μεγάλο τμήμα του ΑΕΠ. ο τουρισμό είναι πάρα πολύ σημαντικό επίση γιατί πρόκειται για μια δραστηριότητα η οποία αφορά και τις νησιωτικές περιοχέ και τι ακτέ ε, καθώς επίσης ε, και απομακρυσμένε ορεινέ περιοχές, δηλαδή όλες αυτές οι περιοχές οι οποίες χρήζουν πραγματικά μεγάλης ανάπτυξης. Ε, για μα, λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να σκύψουμε πάνω στο θέμα του τουρισμού και πρέπει να το κάνουμε πρώτα απ' όλα εστιάζοντας την προσοχή μας σε αυτές τις χώρες, τις περιοχές υποδοχής. Συνειδητοποιούμε βεβαίως ότι υπάρχουν διαφορετικά προβλήματα, έλλειψη ε, ε, νερού, το ανέφερε και η Επιτροπή, αλλά εγώ θα πάω και πιο πέρα ακόμα πιστεύω ότι θα πρέπει να ε, δούμε με ποιο τρόπο μπορούμε να μειώσουμε ενδεχομένως το πώς, πώς μειώνεται το πόσιμο είδο. πώς είναι δυνατόν ας πούμε να ε, ε, επιτρέπουμε να δημιουργηθούν τερέν του γκολφ ή γήπεδα του γκολφ σε περιοχές οι οποίες έχουν ήδη πρόβλημα σε βάση των ερευνών 60% των ε, τουριστικών καταλημάτων στην Ευρώπη ε, εξαρτώνται από την ποιότητα του τουρισμού. Επομένως θα πρέπει να σκύψουμε πάνω στο θέμα αυτό. 80% του διεθνούς ε, τουρισμού γίνεται μέσω από οι οποίες είναι εξαιρετικά επιθετικές για το περιβάλλον και οι οποίες αποτελούν ένα απεπαλαιωμένο σύστημα τουριστικής ανάπτυξης κατά την άποψή μας και θα πρέπει να δούμε, να αλλάξουμε τα πράγματα έτσι ώστε να βελτιωθούν, να είναι θετικά τα αποτελέσματα και για τις ε, ε, περιοχές υποδοχής αλλά κυρίως για περιοχές ε, οι οποίες θα πρέπει περαιτέρω να προστατευτούν λόγω του ότι αποτελούν μια ιδιαίτερη πρόκληση γιατί έχουν ένα ιδιαίτερο φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά κτλ. Επίσης πρέπει να προωθήσουμε μορφές αναλλακτικού τουρισμού και βεβαίω να υπάρξει ισορροπία ανάμεσα στους κοινωνικούς, περιβαλλοντικούς, πολιτιστικούς παράγοντες. Πέραν τούτου, Οπουδήποτε αναπτύχθηκαν εναλλακτικές μορφές τουρισμού έχουν ε, επιτύχει και έχουν ε, επιτύχει επίσης καλύτερη διείσδυση ε, στον τοπικό πληθυσμό αλλά βεβαίως και καλύτερη περιβαλλοντική διατήρηση και προκειμένου υπάρχει περαιτέρω αύξηση του τουριστικού και λοιπού δυναμικού. Περαίνοντας μπορώ να πω ότι οι τομείς όλοι αυτοί του τουρισμού, της ανάπτυξης, της κοινωνίας είναι τομείς οι οποίοι αλληλοσυνδέονται και επομένω θα πρέπει να αναπτύξουμε τον ε, εναλλακτικό τουρισμό έτσι ώστε να έχουμε αρμονική ανάπτυξη καθώ επίση ε, και καλή διατήρηση όλων των περιβαλλοντικών ισορροπιών. Ε, αυτά ήθελα να πω και βεβαίω. θα συμμετάσχουμε και στη συζήτηση κατά τη διάρκεια τη συζητήσεω των τροπολογιών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι αυτή η στρατηγική πολιτική την οποία έχει καθορίσει η ευρωπαϊκή πολιτική μας δίνει καλά μηνύματα, ε, καλά σημάδια όσον αφορά την στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με αυτό την, με αυτόν τον νέο χώρο ανταγωνισμού με τον οποίο ασχολούμεθα. επομένω ε, εκτιμώ την όλη διάθεση. Η γνωμοδότηση ε, Καρόνα είναι εξαντλητική και οπωσδήποτε μπορούμε ε, να μοιραστούμε να συμμεριστούμε τις απόψεις. Θα ήθελα πάντως στα πλαίσια ενός πράγματο εργασίας να υποβάλω κάποιες προτάσεις οι οποίες θα πρέπει να εκλειφθούν ως προτάσεις προς βελτίωση, περαιτέρω βελτίωση των προτάσεων της Επιτροπής. Βεβαίω Ε, να εστιάσουμε την προσοχή μα στην ποιότητα του τουρισμού και στην διαφοροποίηση. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κατά αυτήν τη λογική θα ήθελα να σημειώσω ότι ενδεχομένως αυτός ο προσανατολισμός προς την ποιότητα ε, θα πρέπει να ολοκληρωθεί περισσότερο. Δηλαδή να υπογραμμίσουμε όπως έγινε και σε άλλες επιτροπές ε, την ε, διασύνδεση των πρωτοβουλειών που θα αναλυφθούν έτσι ώστε να ενδυναμωθούν κάποιες ιδιαίτερες μορφές ε, τουρισμού κάτω από την αιγίδα ας πούμε ενός ευρωπαϊκού σήματος που θα αφορά ταυτόχρονα και θα συνδέεται και με την επιστοποίηση των χώρων, των περιοχών σαν ε, περιοχές ε, πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Νομίζω ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει τις ε, περιοχές, διάφορες περιοχές της Ευρώπης. Επίσης, ανάλογα με τις διάφορες μορφές τουρισμού, πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνδέσουμε ε, και τον πολύ σημαντικό δίκτυ που καταθέτει ε, η έκθεση, έτσι ώστε να υπάρξει μεν εκπαίδευση, αλλά να αφορά ε, πιο συγκεκριμένα τις ειδικές μορφές τουρισμού προς ανάπτυξη. Τέλος, Η δράση αυτή είναι πάρα πολύ θετική και είναι σημαντικό κυρίως η δική μας Επιτροπή ε, να είναι ιδιαίτερα προσεκτική έτσι ώστε να μην επιτρέψει η πολιτική του τουρισμού και οτιδήποτε συνδυάζεται με αυτήν να μην λέγω αποσυνδεθεί από την ε, κοινωνική πολιτική και την πολιτική συνοχής. Είναι σημαντική και ικανή αναφορά που γίνεται στο σημείο 3 της γνωμοδότησης, αλλά πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δοθούν και κάποια άλλα μηνύματα πιο αποφασιστικά, πιο ισχυρά. Είναι σημαντικό κατά την άποψή μου να υπάρξει και αναφορά στην ανάγκη που ε, υπάρχει για κάλυψη των ε, αναγκών και των δικαιωμάτων των καταναλωτών. Αναφέρεται κάτι τέτοιο στο σημείο 7, ε, όπου αναφέρεται ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι νέες εξελίξεις και τα νέα εργαλεία που η τεχνολογία μας δίνει, να χρησιμοποιήσουμε τα τεχνολογικά, τις τεχνολογικές καινοτομίες, αλλά ακριβώς πρέπει να προσέξουμε έτσι ώστε να μην έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα σε αυτόν το τόσο ευαίσθητο τομέα. Αυτά ήθελα να πω. Η αναφορά σε μικρές μεσαίες επιχειρήσεις βεβαίως είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι στον τουρισμό η συντριπτικότατη πλειοψηφία αφορά μικρές ή πολύ μικρές επιχειρήσεις και επομένως ε, θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενδεχομένως να αναλάβει στοχευμένες πρωτοβουλίες απέναντι σε αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες χρήζουν ιδιαίτερας προσοχής. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Άλβε, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. Πάρα πολύ σύντομα, κύριε Πρόεδρε. είναι σημαντικό, όπως τονίστηκε, να συμπεριλάβουμε και το φυσικό περιβάλλον μέσα στη στρατηγική του τουρισμού. το δίκτυο Natura 2000 έχει τεράστιες δυνατότητε για να προωθήσει την φυσική ομορφιά σαν στοιχείο του τουρισμού και της διαφοροποίησης. Αυτή είναι η σύντομη λοιπόν παρέμβαση που θέλω να κάνω. Ο εισηγητής θέλει να απαντήσει εν συντομία. Mm, πολύ σύντομα. Για να πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για, την, ε, για τον ουσιαστικό τρόπο με τον οποίο διάβασαν την έκθεσή μου που θεωρώ ε, ότι πραγματεύεται ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Επίσης ε, νομίζω ότι όλα αυτά, όλες αυτές οι παρατηρήσεις και τα σχόλια που άκουσα είναι εξαιρετικά πιστικά και σίγουρα θα, θα τα χρησιμοποιήσω έτσι ώστε να ενδυναμώσω την γνωμοδότηση αυτή. Ε, ε, δεν ξέρω εάν κατάλαβα καλά αυτά που είπε ο κύριος Αγκουράκης αλλά η επιχειρηματολογία ήταν πάρα πολύ απλή λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρώπη είναι ένα από τα ε, ε, ε, ότι η Ευρώπη είναι μια γυραιά ήπειρος, έχει δηλαδή πολλούς <clears throat> προχωρημένης ηλικίας πολίτες. Θεωρούμε ότι ακριβώς ηλικιωμένοι δεν είναι εμπόρευμα, είναι μια νέα δυναμική και επομένως μπορούν να αποτελέσουν μια νέα κινητήρια δύναμη και να κινήσουν στον τουρισμό και να κινήσουν και την οικονομία. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Περιμένω τις τροπολογίες οι οποίες πιστεύω ότι στη συντριπτική τους πλειοψηφία θα γίνουν αποδεκτές γιατί θα ε, ενισχύσουν ακόμα περισσότερο αυτή τη γνωμοδότηση και επομένως ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική εργασία. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Μερσή σε όλους για αυτή την ανταλλαγή απόψε. μόνη απόφαση πρέπει να, κάνουμε, να πάρουμε σήμερα είναι για την προθεσμία τροπολογιών στις 3 Φεβρουαρίου 6 το απόγευμα και τώρα μπορούμε να περάσουμε στο τελευταίο ουσιαστικό σημείο στη μέση διαταξή μας που είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων για, την... για το επιτιβάστο του εγγράφου εργασίας του Μάρκους Πίπερ σε σχέση με την πέμπτη έκθεση συνοχής και της Επιτροπής και θέλω να σας πληροφορήσω ότι είναι μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων. Ο Μάρκους θα παρουσιάσει το κείμενο της έκθεσής του θα έχουμε και πάλι την ευκαιρία να προχωρήσουμε σε μια συζήτηση και θα ήθελα να ζητήσω από τον Μάρκος να κάνει τα εισαγωγικά του σχόλια. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρόκειται, όπως είπατε, για την πέμπτη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Συνοχή και την στρατηγική για την, αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό, για τη στρατηγική για την πολιτική συνοχή με το 2013. Θέλω να εστιάσω σε δύο πράγματα στην έκθεση αυτή. Καταρχήν στην ίδια την έκθεση της Κομισιόν, την πέμπτη έκθεση συνοχής, αλλά και στην ανακοίνωση της Κομισιόν για τα συμπεράσματα τα οποία αντλεί. Αυτά είναι τα δύο βασικά έγγραφα και θα είναι πολύ χρήσιμα αυτά τα οποία έχουν εκπονήσει υπό εκθέσεων οι συνάδελφοι. Η έκθεση του κ. Μιχολάσης για τα διευθυντικά ταμεία 2007 με 2013, η έκθεση Λάστρα για την εφαρμογή της Λισαβόνας και της στρατηγικής Ευρώπη 2020 στην πολιτική συνοχή κτλ. Όπως ε, είπα προηγουμένως, θέλω να εστιάσω πολύ περισσότερο στο μέλλον. Προτού έρθουν οι προτάσεις για τις μελλοντικές προοπτικές, εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν είχαμε μέχρι στιγμής καμία δυνατότητα να εκφράσουμε τη γνώμη μας για τις γενικές κατευθυνσεις της Κομισιόν. Γι' αυτό αυτά τα οποία λέω για το μέλλον περιορίζονται σε ορισμένα μονάχα ζητήματα. Δεν μπορώ να διεξέλθω πιο ειδικευμένα θέματα όπως αυτό το νέο περιφερειακό πλαίσιο το οποίο αναφέρεται ούτε το ζήτημα το οποίο έχει να κάνει με τον στόχο 3. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία πρέπει να τα αντιμετωπίσουν οι επιμέρους εισηγητές. Θέλω να έχω μια διαφορετική τώρα διάρθρωση της έκθεσης από ό,τι διαφαίνεται από το έγγραφο εργασία με την δική σας συνένεση. Μας ενδιαφέρουν τα επιτεύγματα της πολιτικής συνοχής μέχρι το 2010, η, το οικονομικό πλαίσιο και η ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Αυτό πρέπει να είναι το υπόβαθρο και το γενικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε καλύτερα τα θέματα της μελλοντική εξέλιξης της πολιτικής συνοχής και εκεί νομίζω θα πρέπει να δημιουργήσουμε και το μεγαλύτερο χώρο συζήτησης στην Επιτροπή μας. Εκ των προτέρων ορισμένες παρατηρήσεις σε σχέση με αυτά τα οποία προτείνει η Κομισιόν. Κατά την άποψή μου, εδώ και ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, εγώ συμμερίζομαι την άποψη ότι πρέπει να έχουμε μια αντιμετώπιση <clears throat> της πολιτικής συνοχής που να είναι εστραμμένη προς το αποτέλεσμα. Αυτό σημαίνει πρέπει να έχουμε αξιόπιστους δείκτες και μέσα στη στρατηγική της Ευρώπης 2020 έχουμε ήδη μια κατεύθυνση η οποία είναι πιστική αλλά δεν νομίζω ότι θα μπορέσει η Ευρώπη 2020 να καλύψει όλες τις απαιτήσεις μιας πολιτικής συνοχής. Το ίδιο ισχύει σε σχέση με την ε, μελλοντική περιφερειακή πολιτική να εξασφαλίσουμε την υπεύθυνη δέσμευση των κρατών μελών, ιδίως σε ό,τι αφορά τον έλεγχο των κονδυλίων που αποδίδονται στην περιφερειακή πολιτική. Και εδώ, σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με την Κομισιόν αλλά θα πρέπει να υπάρξουν πιο συγκεκριμένες προτάσεις εφαρμογής που να μπορούν να συλλέξουν τη συνένεση και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κρατών μελών. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για όλους μας, η οποία μέχρι στιγμής δεν έχει καλυφθεί πλήρως, δεν έχουμε καταφέρει να καθορίσουμε σαφέστερα τι ακριβώς σημαίνει η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία και τι ρόλο παίζει στην περιφερειακή πολιτική. Και επίσης είναι σημαντικό να υπογραμμίσω αυτό που είπαμε ήδη μέχρι στιγμής για τους ε, δείκτες. Όλα αυτά τα οποία έχουμε μέχρι στιγμής είναι θεωρητικού χαρακτήρα. Πρέπει να πιέσουμε την Κομισιόν να γίνει πιο συγκεκριμένη σε σχέση με το σύνολο των δικτών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν την καταμέτρηση των επιτυχιών. Για την ερεσιμότητα επίσης και για τι εταιρικέ σχέσει με στόχο στην ανάπτυξη. Αυτά που λέει η Κομισιόν είναι καλόδεκτα, αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ θεωρητικά και πρέπει να είμαστε λίγο πιο σαφεί. Εγώ ανησυχώ ιδιαίτερα για το γεγονό ότι αυτή η έννοια τη εταιρική σχέση ε, ανάπτυξης αφορά κυρίω τη συμμετοχή των κρατών μελών. Πώς θα καταφέρουμε όμως οι περιφέρειες να μπορέσουν αυτόνομα και δεσμευτικά να συμμετέχουν σε αυτές τις διαδικασίες εταιρικής σχέσης για την ε, ανάπτυξη. Πρέπει λοιπόν να δούμε καλύτερα μια κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης, κρατών, μελών και περιφερειών που θα είναι αποφασιστική για το μέλλον της πολιτικής ε, συνοχής. Θέτω 36 ερωτήματα, ίσως είναι πολλά, ίσως είναι πολύ φιλόδοξο να περιμένει κανείς να τα απαντήσει κανείς όλα. Ένα κύριος άξονας είναι η στρατηγική Ευρώπη 2020 όπου και εγώ θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αυτή η στρατηγική έχει ορισμένες εγκάσεις οριζόντιες αρμοδιότητες και έχει σαν στόχο να εντάξει την ε, πολιτική συνοχή σε ένα πλαίσιο. Αλλά το να θέσουμε την πολιτική αυτή μόνο στο στόχο της αηφορίας, εμένα δεν μου φαίνεται ότι είναι ικανοποιητικό και δεν καλύπτει όλους τους στόχους μας. Σε επίπεδο προϋπολογισμού τα πράγματα δεν έχουν πάει τόσο άσχημα και οι επιτυχίες στο χρονικό διάστημα 2007-2013 θα πρέπει να μας εταρρύνουν να έχουμε μια καλύτερη ε, εστίαση στο χρονικό διάστημα προγραμματισμού 7 ετών. Για τη στρατηγική 2020 επίσης έχω κάποιες ανησυχίες γιατί τα θέματα της υποδομής, προστασίας του περιβάλλοντος, καινοτομίας ε, και κλιματικής αλλαγής για αυτά συμφωνώ 100%. Αλλά θέτω και το ερώτημα. Πώς θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σε μερικούς κεντρικούς στόχους. Παραδείγματος χάρη να μειώσουμε το ποσοστό αυτών οι οποίοι δεν τελειώνουν το γυμνάσιο και το Λύκειο. Εδώ πρέπει να έχουμε καλύτερη αντιμετώπιση. Πώς θα αντιμετωπίσουμε την ε, ένδυα και τον αποκλεισμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Επίσης θα πρέπει να δούμε τι χαρακτήρα ε, υποδειγματικό παίζει πολιτική συνοχής και να αντιμετωπίσουμε μέσα σε αυτήν και το θέμα της πολιτικής της κοινωνικής. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η Ευρώπη. Μπορεί να φτάσει μέχρι στο κοινωνικό ιστό, στις κοινωνικές ενώσεις, πολιτών, στα σχολεία κτλ. Και γι' αυτό εγώ δεν είμαι απόλυτα σύμφωνος με τη στρατηγική 2020. Πρέπει να είναι σαφέστερη η κατανομή αρμοδιοτήτων μέσα στα πλαίσια αυτής της στρατηγικής. Γιατί ακόμα και αν αποτυγχάνει, αν είναι σαφές ότι αν αποτυγχάνει ένα κράτος στη σχολική του πολιτική, υπάρχουν επιπτώσεις οι οποίες θα έχουν επιπτώσει σε εθνικό επίπεδο. Μπορεί να αλλάξει κυβέρνηση, μπορεί να αλλάξει τη δομή του εκεί. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο όμως πρέπει να το αναλάβει στην δική της ευθύνη η Ευρώπη, σαν σύνολο. Επίσης, θα πρέπει, όπως ελέγχθηκε με τον κύριο Επίτροπο, τα θέματα τα οποία επιλέγουν οι περιφέρειες ω προτεραιότητα θα πρέπει να είναι στη δική του αρμοδιότητα. Επομένω, η πολιτική της Ευρώπης 2020 είναι υπερβολικά πράσινη, αν θέλετε. Συγγνώμη, κυρία Σρέτερ. Θα πρέπει να ξέρουμε ότι το θέμα της ενέργειας δεν είναι μονάχα το θέμα της πράσινης ενέργειας. Θα πρέπει να εξασφαλίσουμε μια σωστή ε, εξασφάλιση πόρων ενεργειακών. Δεν πρόκειται μοναχα λοιπόν για την πρασινοποίηση της Ευρώπης, πρόκειται για καλύτερη σύνδεση των υποδομών μεταφορών, μια καλύτερη χρησιμοποίηση των προγραμμάτων 10-10 για να έχουμε ένα καλύτερο ιστό μεταφορών και θα πρέπει να βοηθήσουμε και τις, περι... τις υπόλοιπε περιφέρειες της Ευρώπης να, να ενταχθούν σε αυτό το πλαίσιο. Όλα αυτά είναι πολύ ενδιαφέροντα ερωτήματα. Υπάρχουν και κάποια τεχνικού χαρακτήρα τα οποία έχω αναφέρει στο έγγραφο εργασία. Θα αναφέρω εν κατακλείδη μερικά από αυτά το θέμα της μείωσης της γραφειοκρατίας στους δημοσιονομικούς ελέγχους, το θέμα της χρήσης ως δείκτη του ΑΕΠ, αν μπορούμε να έχουμε ένα διαφορετικό ε, δείκτη, το θέμα των ενδιαμέσων κατηγοριών, όπως μας το παρουσίασε και ο κ Επίτροπος, είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε πρέπει να το αντιμετωπίσουμε χωρίς να δημιουργήσουμε πρόσθετες πολλαπλές κατηγορίες. Επίσης, έχω και κάποιες, ε, κάποια κριτική στάση για το θέμα των επιδοτήσεων προς τις επιχειρήσεις. Και επίσης, δεν θέλω να μιλήσω για μια συγχώνευση των ε, ταμείων που ασχολούνται με τα θέματα συνοχής, αλλά ίσως μια καλύτερη συνεργασία μεταξύ του Ταμείου ε, Παγκοσμιοποίησης, αντιμετωπίσης των συνεπειών της παγκοσμιοποίησης, με το Κοινωνικό Ταμείο. Και επίσης το θέμα της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να έχει συνέπειες στο, στον χώρο της ε, πολιτικής συνοχής θα πρέπει και εκεί να σκεφτούμε ποιες είναι οι συνέπειε οι οποίες θα προκύψουν σε μια τέτοια περίπτωση ε, διότι και οι δομές των ε, χωρών οι οποίε θα εισέλθουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ληφθούν υπόψη στην πολιτική. Τέλος, το θέμα της χρηματοδότηση. Βλέπετε, αγαπητοί συναδελφοί, ότι έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα σε ψηλό επίπεδο, αλλά με διαφορετικές απόψεις, χωρίς να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση ως Κοινοβούλιο. Εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κληθούμε να συναποφασίσουμε για ένα μεγάλο αριθμό τέτοιων θεμάτων. Θα μπορέσουμε να έχουμε μια ουσιαστική συνεισφορά αν εξασφαλίσουμε τη συνένεση στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου. Θέλω λοιπόν να προσπαθήσω να διερευνήσω δυνατές συμβιβαστικές λύσεις για πάρα πολλά από αυτά τα θέματα τα οποία ανέφερα και χαίρομαι ήδη εκ των προτέρων για τη συζήτηση η οποία θα λάβει η χώρα για τα θέματα αυτά. Η, η Επιτροπή Απασχόλησης βάσει του άρθρου 50, δηλαδή ως συνδεδεμένη επιτροπή θα παίξει και κάποιο ρόλο στα ζητήματα αυτά της ε, συνοχής. Εμείς από τη δική μας πλευρά θα πρέπει να κρατήσουμε όμως τη διάσταση την περιφερειακή, να μην αφήσουμε να περάσει σε άλλες επιτροπές. Γι' αυτό εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε ορισμένα κέρια θέματα. Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, 21-22 Μαρτίου θα έχουμε μια ειδική ακρόαση για το θέμα αυτό της έκθεσής μου. 12 Απριλίου θα υπάρχει το έγγραφο του σχεδίου έκθεσης, θα έπρεπε τουλάχιστον να είναι έτσι σύμφωνα με το πρόγραμμα και τη βδομάδα 9 με 12 Μαΐου θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας και το σχέδιο είναι να έρθει στην Ολομέλεια η έκθεση αυτή τον Ιούνιο. Θα ακούσω τώρα με μεγάλη προσοχή τις ε, προτάσεις σας και ελπίζω σε μια καλή συνεργασία στους επόμενους μήνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ Μάρκους. Σκιώδης θέλουν να το λόγο. George. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχήν τον εισηγητή για την πολύ εξαιρετική και αναλυτική ανάλυση που έχει κάνει στο έγγραφό του. Το έγγραφο εργασίας αποτελεί μια πολύ καλή βάση για συζήτηση, καθορίζοντας ήδη τα κύρια σημεία επί των οποίων επιτρέπει να εργαστούμε στο πλαίσιο της έκθεσης, όπως παραδείγματο χάρη συντονισμός μεταξύ επιπέδων διακυβέρνησης και πολιτικών, συνέργεια ταμείων, συγκέντρωση των πόρων, απλοποίηση, αλληλεπιδράσεις, πώληση πέθρου κλπ. Υπάρχουν ωστόσο άλλα σημεία στα οποία πιστεύω ότι θα εκφραστούν πολύ διαφορετικές απόψεις και συνεπώς θα πρέπει να τα εξετάσουμε λεπτομερώς. Θα ήθελα απλώς να αναφέρω μερικά μεταξύ άλλων. Η εξάρτηση της αποταμίευσης κονδυλίων συνοχής από μακροοικονομικές προϋποθέσεις και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις η διαφοροποίηση και το ύψος της ε, συγχρηματοδότησης, η ενδιάμεση στήριξη, οι μακροπεριφέρειες και πολιτική γειτονίας, η όρη λειτουργίας του αποθεματικού επίδοσης, η διάρκεια της προγραμματικής περίοδου, οι αιτήσιες δηλώσεις διαχείρισης και η διάρκεια της ε, προγραμματικής και η διάρκεια επίσης της προγραμματικής περίοδου. Αυτά και σας ευχαριστώ. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ τον εισηγητή για την εργασία του. Πρόκειται για ένα ποιοτικό έγγραφο το οποίο μας χρησιμεύει ως βάση στις συζητήσεις μας και είμαι βεβαία πως η έκθεση αυτή θα έχει μεγάλη σημασία για την απάντηση σε κάποια από τα ερωτήματα που έχουμε και ως εκ τούτου την υποστηρίζω αμέριστα την έκθεση. Θα πρέπει να δούμε πώς θα μπορούμε να εκπληρώσουμε τους στόχους της στρατηγικής 2020 με τα κονδύλια τα οποία διαθέτουμε, τα ταμεία που έχουμε στην διάθεσή μας. Έχουμε μια πολιτική η οποία λαμβάνει υπόψη όλες τις ε, περιοχές που αντιμετωπίζουν ε, δυσκολίες. Είδα ότι ε, τονίσατε μάλλον σήμερα την προσθέμενη αξία της Ευρώπης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και η Επιτροπή μας χρειάζεται να λάβει υπόψη της αυτήν την προσθέμενη αξία της ευρωπαϊκής πολιτικής. Στο έγγραφο εργασίας ε, τονίζεται ζητήματα που άπτονται της έρευνας, ε, της ανάπτυξης. Αυτό που απαιτείται είναι να βελτιωθεί όλη η δομή, όλη υποδομή της στον τομέα της έρευνας. Δεν αρκεί να επενδύουμε πόρους ε, για την ε, έρευνα και την ανάπτυξη, χρειάζεται οι δομέ ε, να είναι προσαρμοσμένε κατάλληλα στι συνθήκε που επικρατούν σε κάθε κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Παράλληλα, χρειάζεται να υπάρξει μια συνεργασία και ένα συντονισμό με τα ερευνητικά προγράμματα αλλά και τα προγράμματα τα οποία έχουν αναλάβει οι περιφέρειες. Στην χώρα μου, παραδείγματος τη Φιλανδία, πολλά απομένουν να γίνουν πάνω στο ζήτημα. Αυτό έχει τη σημασία του αν θέλουμε να έχουμε αυτά αποτελέσματα. Τώρα, σε ό,τι φορά την καινοτομία, χρειάζονται να ληφθούν και εδώ μέτρα βελτίωση των γνώσεων. Η καινοτομία συχνά παραμερίζεται στο πλαίσιο της συζήτησης αυτής και η Ευρώπη χρειάζεται να κάνει πολλά ώστε να μπορέσει να βάλει στην αγορά τα αποτελέσματα των καινοτομίων μας. Αυτό στις πολιτείες λειτουργεί αποτελεσματικά. Αυτές οι καινοτομίες ε, θα πρέπει να μπορούν να υλοποιούνται στην πράξη με την ε, πρόθεσή τους στην αγορά επίσης ε, αναφέρεστε στο έγγραφο εργασία τα προγράμματα συνεργασίας και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο χρειάζεται να εξετάσουμε περαιτέρω για να δούμε κατά πόσο τα προγράμματα NP μπορούν και στο μέλλον να παραμείνουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της μας και να μην αφαιρεθούν από τις αρμοδιοτητές μας. Χρειάζεται παράλληλα να αναρωτηθούμε για την αποτελεσματικότητα αυτών των προγραμμάτων και ενδεχόμενα να την βελτιώσουμε. Πρέπει να δούμε ποια είναι η μακροχρόνια επίπτωση αυτών των προγραμμάτων, διότι τα προγράμματα, όπως ξέρουμε, μπορεί να συνεχίζονται και αφού ολοκληρωθεί η χρηματοδότησή τους. Υπάρχει επίσης και το θέμα των δημογραφικών προκλήσεων. Αναφερθήκατε στις αεροκατοικημένες περιοχές. Αυτό έχει σημασία για τις φτωχές περιοχές, αλλά και για τις ε, πιο πλούσιες ε, περιοχές και παρατηρώ ότι στην έγγραφα εργασίας αναφέρονται κάποια συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα μας επιτρέψουν να βοηθήσουμε την περαιτέρω εξέλιξη αυτών των ε, περιοχών, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου ο πληθυσμός ε, γυράσκει. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κυρία Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Νομίζω ότι το ουσιώδες στην περίπτωση αυτή είναι να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε μια συνένωση όλων αυτών των στοιχείων που μπορεί να προσφέρει η Επιτροπή μας στον τομέα των διαφθορτικών ταμείων και το του Ταμείου Συνοχής. Δεν ξέρω τώρα αν έχει νόημα αυτά τα 36 σημεία να τα παρουσιάσουμε χωρίς να έχουμε μια συνεκτική θέση. Το θέμα της ε, σύνδεσης της πολιτικής συνοχής με την Ευρώπη 2020. Νομίζω ότι η Μαρία Όλμπρετς είχε δώσει μια σαφή απάντηση ποιες πρέπει να είναι η, η διάρθρωση αυτής της πολιτικής. Καταρχήν η Ευρώπη 2020 είναι μια διακυβερνητική πολιτική. Ξέρουμε ότι όλα αυτά θα γίνουν στα πλαίσια της ανοιχτή μεθόδου συνεργασίας. Αυτή είναι η επεξεργασία που γίνεται. Γίνονται προτάσεις από την Κομισιόν και τα κράτη-μέλη αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για την εφαρμογή αυτής της στρατηγικής. Αυτό καλύπτει πάρα πολλούς τομείς όπου η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξαρτάται από τα κράτη-μέλη, διότι δεν έχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ιδιαίτερη αρμοδιότητα ή διότι, εν πάση περιπτώσει, είναι απαραίτητο ο συντονισμό. Ξέρουμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα οποία γίνονται σε διακρατικό επίπεδο μπορούν να έχουν συνεπίσει και για την πολιτική συνοχή. Και ο Γιάνν Όλμπρετ είπε σωστά ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα τροποποιήσει τη δομή του προϋπολογισμού του για να ικανοποιήσει τους στόχους της Ευρώπης 2020. 2020. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα εξασφαλίσουμε κανένα περιβάλλον, κανένα περιεχόμενο σε αυτή τη στρατηγική, αλλά από την άλλη μεριά δεν πρέπει εμείς να τα φορτώσουμε όλα στην Ευρώπη 2020 και να σταματήσουμε τις, ε, τις απαιτήσει που έχουμε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε λοιπόν μια σειρά από διάφορα ταμεία τα οποία έχουν λόγο ύπαρξης. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορούμε αυτά να τα περάσουμε στην Ευρώπη 2020 και να καταργήσουμε όλα αυτά τα συστήματα και τα ταμεία που υπάρχουν. Εγώ νομίζω ότι είναι απαραίτητο να διατηρήσουμε αυτά που έχουμε αυτή τη στιγμή από τις συνθήκες με το ε, περιεχόμενο που τους δίνουν οι συνθήκες. Εμείς έχουμε μία θέληση να υπάρχουν ε, πιο τολμηρά βήματα χρηματοδότησης, να υπάρχουν ταμεία που να καλύπτουν προγράμματα και όχι μονάχα γενικά σχέδια και αυτά τα οποία είπε ο Επίτροπος Χάν σήμερα το πρωί τα υποστηρίζουμε απόλυτα. Θέλω εγώ σε αυτή την έκθεση να είναι πάρα πολύ σαφές σε αυτή την έκθεση Ποιε από τις προτάσεις της Κομισιόν υποστηρίζουμε, πού θέλουμε εμείς να αγωνιστούμε μαζί με την Κομισιόν και να αντιμετωπίσουμε ενδεχομένως τις αντίμαχες θέσεις των κρατών μελών και η Κομισιόν και εμείς είμαστε το, τα ευρωπαϊκά όργανα. Θέλουμε να υπάρξει η συμπερίληψη και η συμφωνία των περιφερειών και αν το, το θέλει η Επιτροπή αυτό θα είναι πάρα πολύ θετικό. Πιστεύω λοιπόν ότι πολλές από τις προτάσεις Κομισιόν είναι θετικές και είναι πραγματικά ισορροπημένες. Αυτό επομένως θα πρέπει να εξέρχεται και από τη δομή της ε, εκθέσεως που να λέει ορίστε αυτά τα οποία βρίσκουμε καλά στην πρόταση της Κομισιόν και τα υποστηρίζουμε και εδώ θέλουμε να επικρίνουμε ή να τροποποιήσουμε τις προτάσεις της Κομισιόν. Αυτές είναι οι δυνατότητες που έχουμε για να επηρεάσουμε τον ε, κανονισμό και να να μας βοηθήσει να εξασφαλίσουμε κάποια ε, συνένεση. Εγώ δεν έχω λοιπόν κανένα πρόβλημα με το περιεχόμενο της έκθεσης του Μάρκος Πίπερ, απλώς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι θα έχουμε τις απαραίτητες πλειοψηφίες στο Κοινοβούλιο και να σκεφτούμε ότι εάν θέλουμε να έχουμε Περιοχέ τη Ευρώπη οι οποίε δεν θα κινδυνεύουν να πλημμυρίσουν στα επόμενα 20 χρόνια χρειαζόμαστε και μια στρατηγική για την αντιμετώπιση τη κλιματική αλλαγή. Δεν πρέπει να αφήσουμε λοιπόν κάποιε περιοχέ έξω από αυτό το πλαίσιο διότι θα αντιμετωπίσουν προβλήματα την κλιματική αλλαγή και δεν θα έχουν καθόλου παραγωγική ικανότητα. Η κλιματική αλλαγή λοιπόν είναι θέμα επιβίωσης για ένα μεγάλο αριθμό παρακτήων περιοχών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και νησιωτικών περιοχών. Υπάρχουν επίσης και στο νότο της Ευρώπης περιοχές οι οποίες ε, ε, πλήττονται από την ξηρασία. Είναι πολλές περιοχές λοιπόν οι οποίες έχουν να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης, το Περιφερειακό Ταμείο έχει δημιουργηθεί ως ένα εργαλείο ad hoc. Ε, εμείς πρέπει να σκεφτούμε λοιπόν για τη διατήρηση εργαλείων τα οποία είχαν χαρακτήρα ad hoc. Εγώ νομίζω ότι μπορούμε πολύ ε, σύντομα να αντιμετωπίσουμε λοιπόν το περιεχόμενο αυτής της έκθεσης. Εγώ νομίζω ότι τα 36 σημεία αυτά θα μπορούσαν να συντονιστούν λίγο καλύτερα για να υπάρχει δυνατότητα της ε, συσφυριλάτησης κοινών θέσεων μεταξύ των πολιτικών ομάδων μέχρι τον Απρέλιο. Νομίζω μπορούμε να κάνουμε μια πιο έντονη επεξεργασία αυτών των 36 σημείων και ελπίζω και ότι ο συγητής με τους κυριότερους συγητές θα κάνει κάτι τέτοιο. Uh, uh, Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι σε γενικές ε, γραμμές συμφωνήσαμε με τις ε, κατευθύνσεις ε, της <clears throat> τελευταία έκθεση για τι περιφέρειες. Τώρα χρειαζόμαστε λίγο περισσότερο συντονισμό και νομίζω ότι η έκθεση αυτή προ αυτή την κατεύθυνση προχωρεί και συμβάλλει μάλιστα στην ε, συζήτηση. Βεβαίω θέλουμε κίνητρα και λοιπά, θα το έχουμε πει. Υπάρχει ένα σημείο το οποίο θα ήθελα να θίξω τη στιγμή που μιλάμε για υποδομές και χαίρομαι που ο εισηγητής αναφέρθηκε σε αυτό, ξέρουμε ότι στο παρόν ε, πρόγραμμα 75% ε, των, ε, της χρηματοδότησης αναφορά την ατζέντα της Λισαβόνας, κατάρτιση κτλ. Δεν αφήνει επομένως κατά την άποψή μου σημαντικό χώρο για τις υποδομές ενώ γνωρίζομαι πάρα πολύ καλά ότι υπάρχει ακόμα πολύ μεγάλο τμήμα των υποδομών, μεταφορών κτλ. που θα πρέπει να ολοκληρωθεί. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ενεργήσουμε με τρόπο ώστε να υπάρξουν αρκετοί πόροι για τη χρηματοδότηση των ε, υποδομών. Ε, ε, τομείς παρέμβαση και ποσοστά παρέμβαση ξέρουμε, βλέπουμε στο Ηνωμένο Βασίλειο ότι οι περικοπές των δαπανών είναι εξαιρετικά μεγάλε και επομένω θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρξει, να διασφαλιστεί μάλλον η συγχρηματοδότηση. Ε, επομένως για τα επόμενα χρόνια ίσως το πρώτο τμήμα των ε, επόμενων δημοσιονομικών προοπτικών ε, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να βοηθήσουμε ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας στις περιφέρειές μας. Τρίτο σημείο αναφέρεται στη σελίδα 5 της εκθέσεως είναι ο ρόλος των τοπικών αρχών. Οι τοπικές αρχές παίζουν εξαιρετικά μεγάλο ρόλο ε, στην προκειμένη περίπτωση. Θα πρέπει να σιγουρευτούμε ότι οι τοπικές αρχές συμμετέχουν ενεργά στις όλες ε, διαδικασίες ε, να, υπάρχουν και εκ των προτέρων συμφωνίες και συζητήσεις ε, για την ανάπτυξη, αναπτυξιακά προγράμματα. Βεβαίως οι τοπικοί άρχοντες θα πρέπει να ε, έχουν σημαντικό λόγο στην κατάρτιση των προτεραιοτήτων για την κάθε περιφέρεια. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Αγκουράκης παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. νομίζω ότι η έκθεση του κυρίου Πίπερ μας δίνει τη δυνατότητα πραγματικά να πάμε κάπως σε βάθος αυτή τη συζήτηση για, τα, για τους στόχους και το περιεχόμενο της, της πολιτικής συνοχής. Η ερώτησή μου στον ε, κύριο Πίπερ είναι η εξής συγκεκριμένη. Διαβάζω στη σελίδα 3 ότι είναι της άποψης ότι η ελεύθερη διακίνηση ατόμων και η, ε, γενικά η ελεύθερη αγορά δυνητικά ε, εξαλείφθη τα, τις ανισότητες μεταξύ των περιφερειών tendenziell ausgleichen äh, zwischen den äh, Regionen. Το, θέμα το ερώτημα που έχω εγώ είναι το εξής. Ο κύριος ε, εισηγητής λέει ότι κατά την άποψή του αυτές οι ανισότητες εξαλείφθονται μέσω της ενιαίας αγοράς. Άρα και ο ίδιος δεν είναι απόλυτα βέβαιος για το ότι η ενιαία αγορά από μόνη της εξαλείφθη τις ανισότητες που υπάρχουν μεταξύ των περιφερειών και των χωρών. Αλλιώς γιατί να πει κατά την άποψή του. Ε, έχω πραγματικά ένα μεγάλο ερώτημα στο ζήτημα αυτό. Θα ήθελα να σας παραπέμψω και στην έκθεση του κυρίου Μικόλαση, την οποία την ε, ε, συζητήσαμε και την ψηφίσαμε, όπου και ο ίδιος ο κύριος Μικόλασικ λέει ότι εκφράζει την λύπη του για το ότι μόνο 19 χώρες έχουν δώσει όλα τα στοιχεία που έχουν σχέση με το Ταμείο Συνοχής. Μήπως θα έπρεπε να επεξεργαστούμε αυτά τα 19 στοιχεία για να δούμε αν τελικά υπάρχει σύγκληση ή δεν υπάρχει ή σε τι βαθμό υπάρχει. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι το εξή. Επειδή γίνεται πάλι λόγος πολύ για τη στρατηγική 2020 και επειδή κατά τη γνώμη μου η στρατηγική 2020 το μόνο που θα κάνει είναι να αυξήσει τις ανισότητες και όχι να τις ε, μειώσει. Η ερώτηση μου είναι η εξή. Είναι τόσο δύσκολο να κάνουμε μια προσωμείωση, να αναθέσουμε σε κάποιον, να κάνει μια προσωμείωση στις 271 περιοχές της Ένωσης, να εφαρμόσουν τα κριτήρια της ε, Ευρώπης 2020 και να δούμε τι θα προκύψει. Χωρίς να υπάρχουν τα περιφερειακά ταμεία. Τι θα προκύψει. Θα προκύψει σύγκληση ή θα προκύψει απόκληση. Και δεν είναι τόσο δύσκολο να το κάνουμε αυτό το πράγμα και μετά να δούμε τα περιφερειακά προγράμματα τα οποία κατά τη γνώμη μου έχουν νόημα μόνον για να διορθώσουν τις αποκλίσεις που προκαλούν αυτές οι στρατηγικές επιλογές. Το ίδιο έγινε με την στρατηγική της Λισαβόνας, γι' αυτό δεν έχουμε καμία ανάλυση τι έγινε. Το ίδιο θα γίνει και με το 2020, γι' αυτό ζητάω να γίνει αυτή η προσωμείωση και να δούμε ποιο είναι το αποτέλεσμα. Και μετά να δείτε τι ποσά χρειαζόμαστε για να ισορροπήσουμε τις διαφορές. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Ντόιτς. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσω τον κύριο Πίπερ για την εξαίρετη εργασία του. Κάνατε λοιπόν, εκπονήσατε ένα καλό έγγραφο, ε, το οποίο περιέχει πολλά ενδιαφέροντα σημεία. Ε, υπάρχουν βέβαια κάποια με τα οποία δεν συμφωνώ, αλλά δεν έχει έννοια τώρα να σας πω ε, με ποια συμφωνώ, με ποια διαφωνώ. Εγώ θα ήθελα πιο πολύ να επικεντρώσω την προσοχή μου στην μεθοδολογία εργασίας. Πιστεύω ότι η μεθοδολογία που προτείνεται είναι εξαιρετική. Αυτά τα ερωτήματα είναι πολύ ενδιαφέρουσα ιδέα και μάλιστα τα ερωτήματα αυτά είναι πάρα πολύ σοβαρά. Ε, άλλωστε είστε ένας σοβαρός ε, άνθρωπος και επομένως ε, και η ε, μέθοδός σας είναι ε, σοφή, ορθή και σοβαρή. Θα απαντήσω λοιπόν εγώ γραπτά στα ερωτήματα και συστήνω στους συναδέλφους μου να πράξουν ε, ομοίως, να δεχτούν λοιπόν αυτή τη μεθοδολογία εργασίας και να απαντήσουν στα ερωτήματα. Βεβαίως ο Μάρκος θα έχει πάρα, πολύ, ε, πάρα πολλά σελίδες να διαβάζει, αλλά παρόλα αυτά πιστεύω ότι αφού αυτός ξεκίνησε τη διαδικασία με ευχαρίστηση θα διαβάσει όλες αυτές τις απαντήσεις. Έχοντας και τις γραπτές μας ε, απαντήσεις, θα, θα, καταλάβει καλύτερα τις ε, θέσεις μας, ε, θα καταλάβει τι θέλουμε και επομένως ε, θα, γίνει κατά κάποιο, θα αποτελέσει κατά κάποιο τρόπο την, μια προεργασία σημαντική. Δηλαδή θα δει ποια είναι τα σημεία με τα οποία οι περισσότεροι δεν συμφωνούν και θα τα έχει γραπτά μάλιστα, θα τα βλέπει, θα τα θυμάται. και μπορεί να καταρτήσει ένα κατάλογο ε, των ε, ε, ερωτημάτων, των θεμάτων επί των οποίων υπάρχει συνένεση και έναν άλλο κατάλογο με τα σημεία επί των οποίων δεν συμφωνούμε. Αυτά. Πρόεδρος. Ελπίζω ότι δεν θα έχουν όλοι στην Επιτροπή τη Σοφή Λαμπρή ιδέα να απαντήσουν στα ερωτήματα, αλλά εν πάση περιπτώσει, όπως είπε και ο Μάρκος Μπίπερ, θα έχουμε την ακρόαση, θα έχουμε τη συζήτηση της έκθεσης, θα έχουμε την ε, δυνατότητα στους επερχόμενους μήνες να έχουμε πολλή συζήτηση πριν την τελική ψηφοφορία. Αλλά φαντάζομαι ότι ο Μάρκους ε, θέλει να απαντήσει, για να απαντήσει σε ορισμένα από τα θέματα τα οποία εφήγησαν και ελπίζω να μην μακρηγορήσει προβολικά. Αυτή είναι μια πρώτη συζήτηση. Καταρχήν να σας ευχαριστήσω για την καταρχήν υποστήριξή σας. Στον κύριο Σταυρακάκη να πω πως ο συντονισμός των διαφόρων επιπέδων θα αποτελέσει ε, προτεραιότητα. Τις ε, μακροπεριφέρειες θα είναι ένα ζήτημα που θα χρειαστεί να εξετάσουμε και σχετικά με τις περιφέρειες αυτές. Είναι προφανές ότι κατά τη διάρκεια <clears throat> της περίοδου προγραμματισμού το θέμα αυτό είναι καλυμμένο. Ένα άλλο σημείο το οποίο είναι σημαντικό είναι το θέμα της πολιτικής έρευνας με τα, το οποίο θα πρέπει να συνεργαστεί να, με τα προγράμματα τα οποία έχουν διαχρονικό χαρακτήρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα επίσης για την υποστήριξη που δόθηκε από, το εργαλείο, από την ΕΠΑ, από το εργαλείο το προενταξιακό, το οποίο μπορεί να παίξει μεγάλο ρόλο στη δημιουργία ικανοτήτων σε περιφερειακό επίπεδο και επίσης κατανοώ αυτό που το οποίο είπατε ότι πρέπει το δημογραφικό θέμα να είναι πιο σημαντικό μέσα στην έκθεση. Για την κυρία Σουέντερ πρέπει να πω ότι δεν θεώρησα ότι ήθελα να θολώσω τα νερά με το να θέσω τόσα πολλά σημεία. Νομίζω ότι ο στόχος μου είναι να εστιάσω στο μέλλον και δεν έχω κάνει καμία προσπάθεια να θέσω όλα τα θέματα στο μέλλον, δεν το έκανα αυτό. Νομίζω ότι ούτως ή άλλως θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα ζητήματα και το θέμα της ε, κλιματικής αλλαγής. Προφανώς και εγώ δεν θέλω να υπάρξει κάποια ε, να πλημμυρίσουν οι ευρωπαϊκές ε, περιφέρειες και να βρεθούν κάτω από το νερό, αλλά δεν θέλω να δημιουργήσω και πανικό κιόλας για το ζήτημα αυτό. και για το θέμα που έθεσε ο κύριος Σαγκουράκη για τις βάσεις της ενιαίας αγορά. Είναι γενικό ότι η ενιαία αγορά είναι και η βάση για την οικονομική ανάπτυξη, είναι το βασικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μας ε, βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και οι περισσότερες περιοχές της Ευρώπης έχουν καταφέρει να πραγματοποιήσουν αυτή την ανάπτυξη μπορούμε να εξετάσουμε και τις μελέτες κατά περιοχές. Εγώ έκανα οικονομική γεωγραφία στο Πανεπιστήμιο και πράγματι πιστεύω ότι χωρίς την οικονομική ανάπτυξη δεν μπορούμε να έχουμε ούτε προστασία του περιβάλλοντος ούτε περιφερειακή ανάπτυξη. Πρέπει όμως να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει και κάποια σύγκληση των φτωχότερων περιοχών με τις, με τις πλουσιότερες περιοχές της Ευρώπης και επίση ότι όλα αυτά τα οποία θα κάνουν στο περιφερειακό επίπεδο θα συνάδουν με τις προσπάθειες Ευρώπη για τον τομέα τη ενέργεια, τον τομέα τη κλιματική αλλαγή κτλ. Το... Η Ευρώπη 2020 είναι ακριβώς ο τομέας εκεί όπου είναι απαραίτητο να έχουμε δείκτες για να καταλάβουμε τι έχει επιτευχθεί. Θα πρέπει να δούμε ποια είναι τώρα η κατάσταση, ποια θα είναι η κατάσταση σε πέντε χρόνια, τι θα έχουν επιτύχει οι περιφέρειες της Ευρώπης βάσει της περιφερειακής πολιτικής και πρέπει η Κομισιόν να μας δώσει βασικές λύσεις και για αυτό το θέμα. Για τον κύριο Ντόιτσο επίσης θέλω να τον ευχαριστήσω. Νομίζω ότι μπορούμε να έχουμε κοινή γνώμη για όλα αυτά τα θέματα. Αν ανοίγει δηλαδή μια δυνατότητα θα πρέπει να την χρησιμοποιήσουμε όλοι. Όταν φτάσουμε τώρα στο να συγκεντρωθούμε για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε 10 ή 15 μονάχα σημεία από αυτά τα 36 που ανέφερα, αυτό θα είναι θετικό πολιτική άποψη και έχει δίκιο η κυρία Σρέντερ. Εγώ θέλω σε τελική ανάλυση να υποστηρίξω την Κομισιόν στην προσπάθειά τη και να δώσω έμφαση στα σημεία αυτά τα οποία είναι τα πιο σημαντικά. Να πούμε ότι σε αυτά τα σημεία μπορούμε να σα υποστηρίξουμε. Εδώ δεν μπορούμε να συμπορευτούμε μαζί σα και εδώ το Κοινοβούλιο έχει διαφορετικέ απόψει. Έτσι θα μπορούμε να έχουμε μια μεγαλύτερη σαφήνεια στην έκθεση αυτή. Ε, σε ευχαριστώ Μάρκο Πίπερ για την ε, συμβολή σου στην σημερινή συζήτηση. Ελπίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα η μελλοντική συζήτηση. Θα ήθελα τα επόμενα λεφτά που μας έχουν απομείνει να αναφερθώ στις αποφάσεις που έλαβαν οι πολιτικοί συντονιστές. Να σας ενημερώσω πώς λάβαμε απόφαση για την ανάθεση των ε, παρακάτω εκθέσεων και γνωμοδοτήσεων για τις εξαιρέσεις ε, και λοιπά δόθηκε στην Άλντε το προβλήμα του 2012 στο ΕΛΚ για το, το Ταμείο Αλληλεγγύης για έξι κράτη-μέλη στην Πρόεδρο. Η Πρόεδρος ε, θα αναλάβει επίσης και την γνωμοδότηση για το Ευρωπαϊκό Σύστημα Περιφερειακών ε, και Εθνικών Λογαριασμών, Σοσιαλιστές ε, και τους ελιστές μάλλον θα αναλάβουν το λόγο της πολιτικής προστασίας και ανθρωπιστικής βοήθειας για τις προτεραιότητες στον τομέα των υποδομών στο ΕΛΚ. Επίσης αποφασίσαμε πως οι συντονιστές μέχρι την Παρασκευή θα στείλουν τις ε, συνεισφορές τους στην επιστολή που προετοιμάζεται και που θα αποσταλεί την Δευτέρα στην ε, ε, διάσκεψη των Προέδρων Επιτροπών για, σε ό,τι αφορά τη συζήτηση του Μαρτίου για τον, στην Ολομέλεια για τον ε, ε, στρατηγική 2020 επίσης ε, Αποφασίστηκε η συνεδρίαση με τα Εθνικά Κοινοβούλια να διεξαχθεί τον Οκτώβριο και το θέμα θα είναι η νομοθεσία και το, στο ζητήματα πολιτικής συνοχής να έχουμε τις συζητήσεις με τους υπουργού ε, συνοχής ε, θα καλέσουμε τον Ρουμάνο πρόεδρο, ε, υπουργό συγγνώμη. Συμφωνήσαμε ότι όταν οι πολιτικές ομάδες αποφασίσουν να υποβάλουν μια προφορική ερώτηση, τότε η γραμματεία θα είναι υποχρεωμένη να ελέγχει τι είναι καλύτερο ή τι είναι εφικτό, να υπάρξει μια, πολιτική, μια ερώτηση από πλευρά πολιτικών ομάδα ή από πλευρά τη Επιτροπή μα. Ε, επίσης θα προωθήσουμε το θέμα της ε, πολιτικής του Δούναβη στην διάσκεψη των Προέδρων. Αποφασίσαμε επίσης ε, το, για το ζήτημα των μη νομοθετικών ε, μη νομοθετικού περιεχομένου εκθέσεων και η Γραμματεία θα ενημερώσει τους συντονιστές και θα αποφασίζουν οι συντονιστές πώς θα ενεργήσουν σχετικά με το ζήτημα. Αυτά ήταν όλα. Θα ήθελα τώρα να κηρύξω το πέρας της συνεδριάσεώς μας. Εκτός αν έχετε κάτι να θίξετε στα διάφορα, θα συναντηθούμε τον Φεβρουάριο και στην έκτακτη συνάντησή μας στο Στασβούργο, θα εξετάσουμε το ζήτημα της εκθέσεως της αντιπροσωπείας που μετέβει στην Ρουμανία. Γεια σας.